Good morning, everyone. As you slowly take your chairs. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, καθίστε. Θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο Ανδρίου Κάκη στην Επιτροπή μας να μας παρουσιάσει την πρόταση για την διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των αξιολογήσεων κινδύνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα που τον Απρίλιο. Παρόλο που βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της επεξεργασίας της πρότασης για την αδιαφάνεια και την ε, βιωσιμότητα στην τροφική αλυσίδα, είμαι βεβαία ότι ο ε, καθέλην αρμόδιος εισηγητής και ισχυώδης θα θέλουν να εργαστούν σκληρά για να βεβαιωθούν ότι όντως θα υπάρξει περισσότερη διαφάνεια με την απόφαση αυτή, με την ε, νομοθεσία αυτή, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έχουμε λάβει σχετικέ ενημερώσει για το όλο θέμα με τον εμβολιασμό και την ηλεκτρονική υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανταπόκριση στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τον εμβολιασμό. Η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη είναι σημαντική και μας ανησυχούν τα ποσοστά και εσάς και εμάς. Ανυπομονούμε για την παρουσίασή σας, Επίτροπε, και την ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Με μεγάλη μου χαρά έχω την ευκαιρία σήμερα να σας μιλήσω. Γιατί ολοκληρώνεται ένας πάρα πολύ σημαντικός μήνας για την διατροφική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη. Αυτό το λέμε το fitness check, το check-up για αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό ε, νόμο. Και επίσης, σήμερα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πράγματα για τον εμβολιασμό, για την διατροφική ασφάλεια, την υγεία και όλα αυτά θα ωφελήσουν τους Ευρωπαίους. Και θα σας πω ποιες είναι οι εξελίξεις να σας ενημερώσω Οπότε να σας πω πρώτα πρώτα τη νέα πρόταση που αφορά την αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού για τα είδη διατροφής της 11ης Τετάρτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη είχαμε την ευκαιρία ώστε να σας ενημερώσω και αυτό θα το συνεχίσω τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Αυτή η νομοθεσία για τα τρόφιμα θεσπίστηκε το 2002 για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε μια σειρά από κρίσεις που αφορούσαν αυτόν τον τομέα. Και είχαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο από την ΕΦΣΑ και λόγω αυτών των μέτρων ε, αποκτήσαμε το πιο στεγανό σύστημα ασφαλείας για τα είδη διατροφής στον κόσμο. Οπότε με αυτόν τον έλεγχο ε, της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η νομοθεσία μας, το fitness check, που τον ολοκληρώσαμε τον Ιάριο του 18, διαπιστώσαμε ότι όλα λειτουργούν εύρυθμα. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε κρίσεις και προβλήματα από καιρού εις καιρών. Και να γιατί εκπονήσαμε αυτήν τη νέα πρόταση. Οπότε τώρα να αναπτύσσεται αυτή η πολιτική για το πώ θα τα βελτιώσουμε όλα αυτά, να έχουμε περισσότερες δυνατότητε, έχουμε μια σειρά συναντήσεων, συζητήσεων για τα διαφορά θέματα και θα θυμάστε την πρόσφατη πρωτοβουλία για την γλυφωσάτη, οπότε και τέθηκε το θέμα μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου στην διατροφική αλυσίδα και πώς θα θωρακιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος. Οπότε η πρότασή μας ε, διαρθρώνεται με τέσσερις άξονες επί τη βάση της εμπειρίας και της ε, πρωτοβουλίας που αναφέραμε. Οι τέσσερι αυτοί άξονε είναι οι εξή. Πρώτα-πρώτα, διαφάνεια στην αξιολόγηση του κινδύνου. Δεύτερον, ποιότητα και αξιοπιστία μελετών. Τρίτον, βιωσιμότητα και διακυβέρνηση του συστήματο τη ΕΦΣΑ. Και τέταρτον, βελτίωση στην ε, επικοινωνία για τον κίνδυνο. Και έχουμε ε, κάνει κάποιου πρακτικές κινήσεις, ούτως ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες επιπτώσεις ε, για κάθε ένα από τους προαναφερθέντες τομείς. Όλα τα δεδομένα για κάποιες εφαρμογές δημοσιοποιούνται επιμελώς, εγκαίρως και σε ηλεκτρονική μορφή εκτός όταν υπάρχουν κάποιο είδους ε, εμπιστευτικές διαβαθμισμένες πληροφορίες. Επίσης, έχουμε και επιστημονικές μελέτες, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία διέπονται από κάποια νομοθεσία. Επίσης, ε, έχουμε κάποιες ε, μελέτες από πλευράς βιομηχανίας και η ΕΦΣΑ παρέχει συμβουλές για το τι πρέπει να γίνει πριν υποβληθεί αίτηση για χορήγηση κάποιας ε, άδειας. Γίνεται κάποιο διαβούλευση και η ΕΦΣΑ έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να προβεί στην αξιολόγηση του κινδύνου. Σε κάποιες εξαιρετικές περιστάσεις η Επιτροπή μπορεί να αναφερθεί στην ΕΦΣΑ και να ζητήσει επιπλέον μελέτες και σε συνεργασία με τα κρατημέλη η Επιτροπή εφαρμόζει ιδιαίτερα αναβαθμισμένους, αυστηρούς ελέγχους ε, των ε, εργαστηρίων που κάνουν αυτές τις ε, μελέτες. Θέλουμε επίση να θωρακίσουμε τη βιωσιμότητα και διακυβέρνηση του κτήματο τη ΕΦΣΑ και τα κρατημέλη εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΦΣΑ σύμφωνα με την κοινή όπως ακριβώς προβλέπει η κοινή προσέγγιση και επίσης έχουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέσσερις εκπροσώπους της ε, κοινωνίας των πολιτών. Και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει ορισμός κάποιων ειδικών επιστημόνων σε αυτά τα επιστημονικά πάνε αυστηρά κριτήρια όσον την αμεροληψία πρόκειται να ισχύσουν και στο μέλλον. Επίσης έτσι αναβαθμίζουμε τις επιστημονικές δυνατότητες της ΕΦΣΑ. Γίνεται καλύτερη συνεργασία με τους εθνικούς επιστημονικούς φορείς. Επίσης θα έχουμε κάποιο είδους καθορισμό στόχων και αρχών για την επικοινωνία για τον κίνδυνο ούτω ώστε οι πληροφορίε να διέπονται από διαφάνεια, να είναι έγκαιρε και ακριβεί. Οπότε επίση θα θεσπιστεί ένα γενικό σχέδιο, πλάνο, πρόγραμμα όσον αφορά αυτή την επικοινωνία για τον κίνδυνο. Θα διευκολυνθούν τα πλέον μέτρα, θα υπάρξει πλέον πρικοδότηση και πριν προχωρήσουμε θέλω να σας τονίσω ότι έχουμε κάποιο είδους στοχοθετημένη αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαίσιο. Ελπίζουμε ότι έτσι θα καλύψουμε την ε, μέρημνα των πολιτών για διαφάνεια, ασφάλεια. Ε, μέχρι τώρα ο, αυτή η γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα έκανε τη δουλειά της, αλλά από τα πάντα επιδέχονται βελτίωση. Θέλουμε επομένω να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα τώρα γιατί κρίσουμε στο μίσο. Οπότε παρακαλώ δώστε προτεραιότητα σε αυτό το φάκελο, σε αυτό το θέμα, ούτω ώστε να ωφεληθούν όσο γίνεται πιο σύντομα οι συμπολίτε μα. Και τώρα, για να δούμε τα θέματα του εμβολιασμού, κύριοι βουλευτέ. Όπω επομένω και ο εμβολιασμό για την Ελλάδα είναι κάτι από τα πιο σημαντικά, ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν και έχουμε 14.000 ε, πρόσωπα τα οποία αρρώστησαν το 2017 τρεις φορές περισσότερο από το 2016, 57 θάνατοι ε, από το 2016, αυτό είναι απαράδεκτο, είναι οδυνηρό. Παρ' όλα αυτά σε όλη την Ευρώπη ο Λένα και περισσότεροι αποφεύγουν τον εμβολιασμό. Γιατί, Γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση από αυτούς που πρεσβεύουν ε, την αποχή από, τη, από τον εμβολιασμό, έχουμε αυτές τις ψευδείς ειδήσει, έχουμε δυσπιστεί από τον κόσμο και επίσης ε, όλοι φοβούνται κάποιο είδους ε, ε, συμπτώματα και παρενέργειες. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς ε, αξιόπιστες πληροφορίες και επίσης υπάρχουν και ελλείψεις στον αφορά τις προμήθειες των εμβολίων και έχουμε στρατευθεί όπως και εσείς τόσο ώστε να λυθεί αυτό το θέμα. Και την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλη εγκρίθηκε ένα σχετικό κείμενο και ένα ψήφισμα και πρόκειτο για την πρόταση για σύσταση από πλευρά του Συμβουλίου και μια ανακοίνωση ούτω ώστε να ενδυναμωθεί η συνεργασία ε, κατά αυτών των ασθενειών που είναι δυνατόν να καταπολεμηθούν με εμβολιασμό. Θα πρέπει να δούμε επίση τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει να υπάρχει αυτού του είδου ε, η, ε, η αποχή από τον ε, εμβολιασμό και να αυξηθεί η η προσέλευση των πολιτών για τον εμβολιασμό, να μπορέσουμε να καλύψουμε τους πιο ευάλωτους, να υπάρχει η ιδέουσα συμβατότητα όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα των εμβολιασμών, να υπάρχει ε, αρκετό απόθεμα εμβολίων, καλύτερη, ε, καλύτερη συνεργασία και επομένως ε, οι επαγγελματίε του κλάδου έχουν σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να ληφθεί μια σειρά μέσων. Θα πρέπει όλη αυτή η πληροφορία να γίνει πράξη όλη αυτή η πρωτοβουλία. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε το ότι αν δεν κάνουμε κάτι τα παιδιά θα συνεχίσουν να πεθαίνουν από τέτοιε ασθένειε που προλαμβάνονται με, την, ε, με τον εμβολιασμό. Ε, αυτό είναι απαράδεκτο και θα συνεχίσουμε να ε, συνεργαζόμαστε και έτσι θα ε, δούμε το, κάτι άλλο. Δηλαδή έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ώστε να ολοκληρώσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά και σχετική στρατηγική και υπάρχει η σχετική ανακοίνωση, αυτή η οποία χθε ε, εγκρίθηκε ούτω ώστε αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν και να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και συστημάτων υγείας των κρατών μελών και έχουμε τρεις άξονες και έτσι θα υπάρξει πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα για την υγεία και ε, με αυτή την ανακοίνωση θέλουμε να υποστηρίξουμε το e-health digital service infrastructure, δηλαδή την υποδομή για, την, για το ψηφιακό σύστημα υγείας. Αυτό είναι δέσμευση των 22. Και έχουμε τώρα το, αυτό το, το, πρόγραμμα ανταλλαγής ε, δεδομένων που αφορούν την υγεία και να έχουμε ακόμα καλύτερη ανταλλαγή δεδομένων. Όλα αυτά θα λάβουν θεσμική επίσημη μορφή, ούτω ώστε οι εργαζόμενοι στην υγεία αλλά και οι ασθενεί να μπορούν διασυνοριακά να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Νέε συσκευέ, τεχνολογίε έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο όγκο τώρα από τέτοια δεδομένα υγείας, τα οποία όμω είναι εδώ και εκεί. Ο δεύτερο πυλώνα σημαίνει ότι πρέπει ε, να διασυνδεθούν όλα αυτά, να συγκεντρωθούν και έτσι να έχουμε ε, ό,τι χρειάζεται η κάθε περίπτωση από πλευράς ε, πρόληψης και αγωγής. Πρώτο βήμα είναι αυτή η δήλωση, διακήρυξη των, των 16 της 10 Απριλίου, ούτω ώστε να έχουμε ένα εκατομμύριο ε, γονιδιώματα και αυτά να είναι προσβασίμα μέχρι το 2022 όσον αφορά τις ε, υπάρχουσες πρωτοβουλίες για μια ιατρική ακριβίας. Τα δίκτυα αναφοράς συλλέγουν τα δεδομένα και υπάρχει και ένα ιντερνετικό σύστημα ε, διαβούλευσης και παροχής ιατρικών συμβουλών. Θέλουμε να υπάρχει κινητή υπηρεσία υγείας, να υπάρχει παροχή ε, συμβουλών από απόσταση νέα μοντέλα φροντίδας και έτσι οι πολίτες να μπορούν να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην ε, φροντίδα της ίδιας τους της ε, υγείας. Με τέτοιες τεχνολογίες επομένως, ε, εάν έχουμε συντονισμό, θα μπορέσουμε να κάνουμε τον τομέα της υγείας ικανό να ωφεληθεί από την ψηφιακή επανάσταση κάποια σχόλια τώρα όσον αφορά την πρόταση αυτορύθμισης που πρόσφατα ε, υπέβαλε η βιομηχανία αλκοολούχων ποτών. Τώρα αξιολογούμε την πρόταση. Αλλά με αυτή την ευκαιρία να σας πω τα βασικά της σημεία. Πρώτα-πρώτα, υπάρχει ένα κομμάτι αυτής της πρότασης που θα αφορά όλον τον κλάδο και θα έχει κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Το άλλο τμήμα της πρότασης έχει ανατομέα κάποια παραρτήματα για μπύρα, αλκοολούχα, κρασί, ε, ε, μιλίτη και κρασί από φρούτα. Και εκεί περιγράφονται κάποιες επίση δεσμεύσεις για κάθε υποτομέα. Θέλουμε να είναι η προσέγγιση σε κάθε τομέα συνεπής με τους άλλους και θα πρέπει να υπάρχει για κάθε εμπορευόμενο ευελιξία. Να παρέχονται πληροφορίες για το τι περιέχει το κάθε ποτό ε, και στην ετικέτα και αλλιώς. Και ανακύπτουν κάποια ερωτήματα ότι θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω η πρόταση, να γίνει τελικά η υλοποίησή της και θα τα ξανασυζητήσουμε στις λεπτομέρειές του τα θέματα, αλλά σας τονίζω ότι είναι σημαντικό να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή την προσπάθεια. με κύριοι βουλευτές, ε, μίλησα διαμακρών σήμερα όσον αφορά αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε ε, τις επιδόσεις μας και στην υγεία και στην διατροφική ασφάλεια για όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει επομένως να συντονιστούμε, θα πρέπει να συνεργαστούμε και εν κατακλείδη έχω να σας πω ότι με την Επιτροπή σας ε, διακαώς επιθυμώ να συνεργαστώ, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για την διατροφική ασφάλεια, να αυξήσουμε την συμμετοχή του κόσμου στους εμβολιασμού και να αυξήσουμε και την εμπιστοσύνη του στα εμβόλια, να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφιακά στην τομέα της υγείας για να ωφεληθούν σε όλη την Ευρώπη οι συμπολίτε μας. Uh, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε, για τα σχόλιά σας σήμερα και να ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο έρωτα από τους συντονιστές. Με δύο λεπτά για κάθε συντονιστή και μετά να ακούσουμε για την υπόλοιπα μέλη στο δεύτερο γύρο έρωτα Ο κύριος Λίζα, ασφαλώς, πρώτος πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Επίτροπο. Και θα ήθελα να δείξω ένα θέμα καταρχάς ένα θέμα το οποίο το ΕΛΚ το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε ένα έγγραφο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Πολύ φιλόδοξη στόχη που έχουμε θέσει. Θέλουμε να συμβάλλουμε κι εμείς ε, το λιθαράκι μας. Δεν μπορεί να τα πετύχει φυσικά όλα η Ευρώπη, αλλά ό,τι μπορούμε να το πετύχουμε προκειμένου σε 20 χρόνια στην Ήπειρό μας να μην υπάρχουν πλέον θάνατοι από καρκίνο. Έχω μιλήσει και με επιστήμονες οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και αν φυσικά και τα κράτη-μέλη συμβάλλουν αυτά που τους αναλογεί. Πολλά λοιπόν στοιχεία υποστηρίζουμε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τη τεχνολογία υγεία. Η κυρία Καμπεσόν είναι η συγγήτρια, προκειμένου αυτή η πρόταση τη Επιτροπή να περάσει το συντομότερο δυνατόν προκειμένου η θεραπεία να φτάσει στον ασθενή και να αναπτύσσουν τελικά μόνο θεραπείες που έχουν όφελος για τον ασθενή. Υπάρχουν και άλλε προτάσει για την καλύτερη δικτύωση, για παράδειγμα των μητρώων καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και περιμένουμε μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την κατεύθυνση αυτή. Μα απασχολεί το θέμα αυτό. Ό,τι μπορούμε εμεί να κάνουμε, να το κάνουμε. Κατά δεύτερον, το θέμα των αντιβιωτικών. Έχει κάνει πάρα πολλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω Κοινοβούλιο, πώ να το κάνουμε. Περιμένουμε κι άλλα. Πιο πολλά. Έχουμε την έκθεση πρωτοβουλία τη Κάριν Κάρνμπαχ και θα ήταν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει το συντομότερο δυνατόν ε, μια πρόταση για το πώ θα πετύχουμε να παράγουμε νέα αντιβιωτικά. Γιατί κάθε εβδομάδα πεθαίνουν άνθρωποι. Γιατί πλέον τα αντιβιωτικά έχουν χάσει την ισχύ του. Αποστήλαμε επιστολή προ τον Πρόεδρο για το ότι δεν συμφωνούμε να σταματήσει να καταθέτει προτάσει από το Μάιο και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να χρειαστεί και το φθινόπωρο να έρθει αυτή η πρόταση. Τέλο. να πω και δύο λόγια για το πρόγραμμα εργασία ε, και το πρόγραμμα δράση για την υγεία. Θέλουμε να υπάρχει ε, αυτόνομο πρόγραμμα, όχι να ενταχθεί σε κάποιο υποπρόγραμμα στην, ε, στα προγράμματα ενιαίας αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίζε και κυρία Κάντμπαχ. Επίτροπε. Πολύ σας ευχαριστούμε για τις δηλώσεις σας. Και όπως πάντα διαπιστώνουμε ότι είσαστε πάρα πολύ δραστηρίους και, δραστηρι... και δεσμευμένους. Οι συνάδελφοι θα κάνουν ε, κάποια σχόλια για τα θέματα που θίξατε για τα εμβόλια, για την βιομηχανία. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Λίζα. Μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε ό,τι αφορά τα προγράμματα 2020-2027 Υπάρχει αυτή η προοπτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει αυτά τα προγράμματα για την υγεία στα προγράμματα ενιαίας αγοράς σε, σε μια υποκατηγορία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ζητούσε φιλόδοξη πολιτική για τη δημόσια υγεία για να συμπληρωθούν οι δράσει των εθνικών κρατών μελών, γιατί αυτό είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστό πρόγραμμα. Αυτό θα διευκολύνει και την αξιολόγηση από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να μπει και πάλι η δημόσια υγεία ως προτεραιότητα και να αποτελέσει στο επόμενο που αυτόνομο πρόγραμμα. Θα έχουμε και εκλογές του χρόνου. Ένα από τα βασικά θέματα στα οποία οι πολίτες έχουν ακόμα εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία στον τομέα της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας, είναι ακριβώς η υγεία. Αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε για το μέλλον. Η δημόσια υγεία θα πρέπει να παραμείνει δημόσια υγεία και όχι να ενταχθεί ως υποτμήμα τη ενιαία αγορά. Ευχαριστώ, ο κ. Πιέκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Να μην ε, επαναλάβω αυτά που ήδη ακούσαμε από τους συναδέλφους και από εσάς. Αλλά κάτι από αυτά που είπατε στο πρώτο τμήμα της παρέμβασής σας ε, με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων. Ως ε, πολίτης και ευρωβουλευτής με τρομάζει η έλλειψη διαφάνειας στον τομέα αυτό. Συμφωνώ με τη γενικότερη ανησυχία σε ό,τι αφορά την διάθεση σημαντικών πληροφοριών προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατείνεται ότι η ΕΦΣΑ και οι σχετικές αξιολογήσεις από πλευρά της ΕΦΣΑ θα δημοσιευτούν και θα δημοσιεύονται σε ένα ειδικό στο χώρο. Στην πραγματικότητα, οι μεγάλες εταιρείε ήδη δραστηριοποιούνται προκειμένου να δημοσιευτούν αυτές οι πληροφορίες, αυτά τα δεδομένα. Παρά αυτά, η Επιτροπή μας λέει ότι κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα θα παραμείνουν απόρριτα. Δεν πρόκειται δηλαδή να διατίθενται σε τρίτα μέρη. Πολύ συχνά για αυτές ακριβώς τις πληροφορίες μιλάμε. Αυτό Αυτές είναι οι ευαίσθητες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Και προφανώς ε, η αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων ενδεχομένω να διακυβεύσει κάποιες εταιρείες. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς θα καταφέρετε να συγκεράσετε αυτά τα δύο αντικρουόμενα συμφέροντα από τη μία την, το δικαίωμα του κοινού να έχει πληροφορίες και από την άλλη την ανάγκη να υπάρχουν ε, απόρριτα στοιχεία. Αυτό ενδεχομένω να οδηγήσει σε μια διευθυντήτητα μεταξύ καταναλωτών και οικονομικού κλάδου και ελπίζω τέτοιε ε, αποφάσεις να μην λαμβάνονται αυθαίρετα. Πείτε μας λοιπόν. Thank you very much. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία ευχαριστώ Πρόεδρε, και ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσία σας σήμερα. Μια ερώτηση που αγγίζει και τα τρία θέματα που αναπτύξατε σήμερα το πρωί. Την ε, διαφάνεια ζωτική σημασία. Η πρόταση που υποβλήθηκε πριν από 15 μέρε από εσά και τον κύριο Τίμερμανς για τη διαφάνεια στα επιστημονικά στοιχεία που ε, κατατίθεται στην ΕΦΣΑ. Θέλετε οπωσδήποτε να συμπληρώσετε αυτό το κενό εάν θέλουμε να καλύψουμε και το χάσμα που μας χωρίζει από τους Ευρωπαίους πολίτες και να ενισχύσουμε την επικοινωνία μας προς αυτούς για τους κινδύνους της τροφικής αλυσίδας. Και μετά μιλήσαμε και για την ενεργό συμμετοχή των εταιριών, εάν θα χρηματοδοτούν και αυτές κάποιες μελέτες. Υποβάλαμε μια ε, σειρά από γενικές ερωτήσεις για το θέμα αυτό, πρώτη στην Επιτροπή. Ας πάμε λίγο παραπέρα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ε, σήμερα το πρωί στη συζήτησή μας για το Για το ghostwriting, για τους ε, ε του ε, τους ανώνυμους ξέρετε, το συζητήσαμε και με το Monsanto Papers και πολλές φορές ανατίθεται μια μελέτη έρευνα ε, σε κάποιον ο οποίος δεν αναλαμβάνει την επωνυμία τη έρευνα. Αυτό το καταδικάζει η επιστημονική κοινότητα, αλλά είναι κάτι που οι εταιρείε το κάνουν πάρα πολύ συχνά. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε στην Ευρώπη για να πάψει αυτή η πρακτική. Ε, και μια ακόμη ερώτηση στην πρότασή σας. Ε, υπάρχει στον κατάλογο που λάβαμε προδεκανθιμέρου. μέρου. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε με την παραγγελία συμπληρωματικών μελετών. Γιατί όμως να την έχει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα να παραγγέλνει τέτοιες μελέτες δεν θα ήταν αποτελεσματικό και καλό να μπορεί και η ΕΦΣΑ ή και τα κάτι μέλη να παραγγέλνουν τις πληρωματικές έρευνες ή μελέτες εφόσον χρειαστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που μας διευκρίνησε ποια θα είναι τα σχέδιά του στο μέλλον. Έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω. Καταρχάς, αμφιβάλλω κάπως σε ό,τι αφορά τα μέτρα που αφορούν την αύξηση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά το γενικότερο δίκαιο για το τρόφιμα. Μια εταιρεία, για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλει να κάνει μια, ένα αίτημα για ζανιεκτών, για πρόσθετα τροφίμων. Πείτε μας, ε, σε ποιες περιπτώσεις θα δώσετε συνένεση για να αντιτηρηθούν ε, απόρριτα κάποια δεδομένα. Γιατί δηλαδή να είναι απόρριτα κάποια στοιχεία. Και κατά δεύτερον, προτείνεται μέτρα για την αύξηση της ποιότητας ε, των μελετών ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις μελέτες επαλήθευσης από πλευρά της ΕΦΣΑ. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι, αυτό τι σημαίνει ότι θα ελέγξουμε και τις ήδη διενεργηθήσεις μελέτες για να τις απελευθεύσουμε ή θα κάνει δικό της, ε, δική της έρευνα από εκεί και πέρα η ΕΦΣΑ. Και μία ερώτηση να κάνω για την ε, εμβολιασμό. Λέτε ότι ο εμβολιασμός είναι ένα μέτρο για να προλάβουμε την αντιμικροβιακή αντοχή. Αλλά οι μεγαλύτερε αιτίε ε, για την αντιμικροβιακή αντοχή είναι η υπερβολική χρήση από τον άνθρωπο και στην κτηνοτροφία. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη μείωση της συντατικής κτηνοτροφίας γιατί αποτελεί μια σημαντική απειλή για την υγεία και επίσης αναφέρεται ότι ο εμβολιασμό των ζώων μπορεί να καταπολεμήσει διασυνοριακές επιζωτίες αλλά Μήπως ήταν πιο αποτελεσματικός τρόπος, μιας και για μερικές ασθένειες δεν υπάρχουν ε, ε, εμβολιασμοί, να αποφύγουμε απλά τις δημιουργικές μεταφορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Χόσλινγκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Επίτροπε, για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας διαφάνειας. Φυσικά και συμφωνούμε με τη γενικότερη αρχή, αλλά ο διάλογος κρύβεται στις λεπτομέρειες πάντα. Το θέμα λοιπόν είναι το πώς το θέμα του απόρριτου ή του επαγγελματικού απόρριτου θα οριστεί. Γιατί πολύ φοβόμαστε ότι κάποιες ε, έρευνες απλά δεν θα δημοσιεύονται από εδώ και πέρα. Και έχουμε και τον κανονισμό για τα φάρμακα, όπου τα πράγματα ρυθμίζονται σχετικά ξεκάθαρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο όμως εδώ. Πάτα θα έχει λοιπόν ε, ε, προτεραιότητα το επιχειρηματικό απόρριτο. Γιατί δεν ακολουθήσατε ακριβώ την ίδια εδώ με τον κανονισμό για τα φάρμακα. Κατά δεύτερον, κατά την ε, καταχώρηση τέτοιων μελετών. Τι θα γίνει αν κάποια στοιχεία δεν τα αποκαλύψουν οι εταιρείε αυτέ στην ΕΦΣΑ. Υπάρχει υποχρέωση τέτοια αποκάλυψη στοιχείων. Και ύστερα στην παρέμβασή σα είπατε ότι η ΕΦΣΑ θα έχει δυνατότητα να κάνει δικέ τη ε, μελέτε και ότι αυτό αποτελεί τμήμα τη πρόταση. Αλλά μίλησατε για έκτακτε καταστάσει και περιστάσει. Ε, τι αποτελεί έκτακτη περίσταση. Έχει τι ανάλογέ εμπειρογνώμονες η ΕΦΣΑ για να κάνει για παράδειγμα δικέ τη μελέτε και έρευνε. Έχει τα χρήματα και ύστερα το θέμα των εμπειρογνωμόνων. Πάντα υπάρχει ένα θέμα, γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς και αρκετοί εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Τι θα κάνετε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή και αυτό φυσικά είναι θέμα χρηματοδότησης στη τελική ανάλυση. Και αν παραμένουν τα κρατήρια τόσο αυστηρά, ε, θα μπορέσουμε να αγγιθούμε τελικά την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων. Και τέλος, ε, είπατε ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται οι μελέτες, αλλά με τρόπο που να είναι μηχανικά ευανάγνωστος, προκειμένου να μπορούν να διαβάσουν και οι πολίτες. Ε, κυρία Ντορνανό, ευχαριστώ Πρόεδρε. κύριε Επίτροπε, θέλω να επανέλθω στη γλυφοζάτη. Έχω απευθύνει πολλές συγκεκριμένε ερωτήσεις στην ΕΦΣΑ στα πλαίσια της ειδική Επιτροπής για τα φυτοφάρμακα, ε, όπου είμαι μέλος και συντονίστρια εκ μέρους της ομάδας μας. Είναι ε, απίστευτες οι απαντήσεις της ΕΦΣΑ. Ε, ναι, εξουσιοδότηση. δεν έγινε σεβαστή από τη Γερμανία, ιδίως για την εξακρίβωση στοιχείων των ερευνών και κυρίως την ακρίβεια των επιστημονικών δεδομένων. Ο κίνδυνος της ενεργού ουσίας από την ΕΦΣΑ δεν έχει γίνει ε, πλήρως και κυρίως η πλαστογραφία από έγγραφα της Μονσάντο, που χρησιμοποίησε η ΕΦΣΑ δεν είναι λέει πλαστογραφία. Επιπλέον ε, η σύγκρουση συμφερόντων ε, στο επίπεδο της ΕΦΣΑ δεν υπάρχει. Η ΕΦΣΑ δεσμεύτηκε τον Ιούνιο του 2016 σε μεταρρύθμιση για να ενισχύσει την ανεξαρτησία των επιστημόνων και της αποσχόλησής της, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα από όλο αυτό. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, ή η ΕΦΣΑ δεν λέει την αλήθεια, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά σοβαρό, διότι αυτή είναι υπεύθυνη για την ε, τροφική ασφάλεια, ή η ΕΦΣΑ λέει την αλήθεια, οπότε αναρωτιόμαστε γιατί το Κοινοβούλιο αποφάσισε να δημιουργήσει ειδική επιτροπή μετά το σκάνδαλο της Monsanto Papers. Κι όμως, κατόπιν της πρωτοβουλίας ε, των πολιτών κατά της γλυφοζάτης και των τοξικών φυτοφαρμάκων, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη διαφάνεια και τον ανεξαρτησία των επιστημονικών μελετών βάσει των οποίων διεξάγονται οι ε, αξιολογήσεις της ΕΦΣΑ και η ίδια της διαχείριση, την εσωτερική διοργάνωση. Δεν σας αφήνει λοιπόν άφωνο η απάντηση της ΕΦΣΑ από τότε που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο είναι προσδοκίες των πολιτών. Πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ως προς την διαφάνεια για θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Thank you very much and, uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Μελά. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θέλω να σας ρωτήσω και εγώ για το πρόβλημα της διαφάνειας όπως όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Η διαφάνεια σε θέματα επιστημιστικής ασφάλειας. Το σχολιάσατε κύριε Επίτροπε και είπατε ότι θέλετε ενισχυμένη συνεργασία με, τη, με τα εθνικά επιστημονικά ιδρύματα. Κατανοητό και απαραίτητο. Το ερώτημα είναι το εξή. Πώς σκοπεύετε να συνεργαστείτε με τις επιστημονικές αρχές χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε με βάση ε, συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Χώρες οι οποίες έχουν ειχνηλασιμότητα στα γεωργικά και εκτιματροφικά τους προϊόντα αλλά κάποιες φορές καμία και μάλιστα είναι αδύνατο να εντοπίσει κανείς την αλυσίδα παραγωγής. Για τα φάρμακα τώρα, ε, η η ο εμβυλιασμος συμφωνα με ενώση με συγκεκριμενες ενωσεις γιατρων δεν ειναι ο τρόπος να αντιμετωπιστουν καποιε μεταδοτικε ασθενειε ε, η καλη υγιεινη και το να πλύνει στα τα χέρια του είναι το σωστό. Πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε κάποιες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που ζουν σε κακές συνθήκες ίσως ή δεν έχουν την ίδια δυνατότητα αντίστασης επειδή είναι ξέρω εγώ μετανάστες. Αλλά να λέμε ότι εμβολιασμό είναι η δεν εχουν την ιδια δυνατοτητα αντιστασης επειδη ειναι ξερω εγω αλλα να λεμε οτι εμβολιασμο ειναι η λυση για όλα είναι πραγματικά ε, ψευδής είδηση θα πρέπει να επανέλθουμε και να το ξαναδούμε, διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι η αντίσταση στα αντιβιωτικά θα αντιμετωπιστεί με εμβολιασμό. Και επίσης ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτείτε και κατά πόσον η ηλεκτρονική υγεία, η ψηφιακή αντιμετώπιση της υγείας δεν θα καταστρέψει τις σχέσεις ε, και την επαφή μεταξύ των ανθρώπων, την αλληλεπίδραση, καθώς και τη σχέση ασθενούς και γιατρών. Και πώς ε, τελικά οι φαρμακευτικές εταιρείες μέσω του γιατρού θα μπορούν να παράσχουν και την κατάλληλη αγωγή. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνει το πρώτος γύρος ερωτήσεων. Αν θέλετε, Επίτροπε, να πάρετε ένα πρώτο πακέτο και να το απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ και να αρχίσουμε με την ερώτησή του του κυρίου Λίζα. Ναι, θα πρέπει ο καρκίνος να είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Έχουμε τώρα την ευκαιρία. Με τον Μουέντας τα συζητούμε και με την άβραση και την ε, Μαρία Γκάμπριελ για να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε από κοινού να έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και με τη βοήθεια της πληροφορικής και των υποδομών όπως τα δίκτυα αναφοράς να δούμε πώς θα φτάσουμε σε κάποιες πλατφόρμες και έτσι η αγωγή και η θεραπεία του καρκίνου να αναβαθμιστεί. Χαίρομαι που είναι η κοινή μας η προσπάθεια. Χαίρομαι που νόσαμε τις δυνάμεις μας. Τώρα έχουμε την προοπτική του του δημοσιονομικού νέου πλαισίου. Οπότε τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα καταφέρουμε στο μέτωπο αυτό. Διάβασα μεγάλη προσοχή το έγγραφό σας. Να δώσουμε νέα μορφή στην έρευνα για αντιμετώπιση του καρκίνου. Τώρα διαμορφώνουμε την πρότασή μας, την παρουσιάζουμε στο Συμβούλιο και ελπίζουμε κάποιες χώρες να τις πείσουμε να μας υποστηρίξουν. Και βέβαια θα πρέπει να πείσουμε τη Γερμανία για να κάνουμε βήματα πρόοδο. Είναι τώρα η σωστή στιγμή, ούτως ώστε τελικά Συμβούλιο να ολοκληρώσει τη σχετική συμφωνία. Και όσον αφορά την τεχνολογική αξιολόγηση, όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2019. Και όσον αφορά τα αντιβιωτικά τώρα, όπως είπαμε, περιμένουμε την μελέτη, η οποία θα ολοκληρωθεί το Μάιο. Και θα συζητήσουμε μετά και θα δούμε τι θα γίνει, τι κίνητρα θα δοθούν για φάρμακα γενικώ, συγκεκριμένα για τα αντιβιωτικά. Αλλά πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ τώρα τα συζητούμε. και κύριε κυρία Κάντενμπαχ, όπως και εσείς μιλήσατε για εκείνο το πρόγραμμα. Και θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε, στις όλες πολιτικές γενικά, αλλά στην κάθε μία χωριστά. Συνεχίζονται τώρα οι επαφές και η συζήτηση, οπότε και το σχετικό πρόγραμμα θα έχει στον προϋπολογισμό ένα δικό του αφιερωμένο κεφάλαιο και σας διαβεβαιώ συμφωνούμε για το πρόγραμμα το ερευνητικό. Και βέβαια θέλουμε να επενδύσουμε ε, και θα το βάλουμε σε αυτό το τομέα το πρόγραμμα, στην επένδυση στον άνθρωπο και όχι στα της ενίας αγοράς. Είναι κοινή η θέση των ε, επιτρόπων γι' αυτό. και για τα προγράμματα υγείας. Επισημαίνω ότι έχουμε πολλά και διαφορετικά προγράμματα στα πλαίσια του οριζόντος 2020 και άρα μπορούμε να επενδύσουμε για θέματα φροντίδας της ε, υγείας. Γενικότερα για την υγεία. Γιατί και στον κοινωνικό πυλώνα τώρα προβλέπεται να καλυφθεί η ιατρική φροντίδα και έχουμε και διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα για τον ίδιο σκοπό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία μέσων. Αλλά βέβαια και θα πρέπει να υπάρχει ένα χωριστό πρόγραμμα και συμφωνώ μαζί σας. Μου μιλήσατε επίσης και για έλλειμμα διαφάνειας και για το πώς μπορούμε να βρούμε εγγυήσει ότι θα υπάρξει μια μελέτη και εμπιστευτικός χαρακτήρα των πραγμάτων θα αναδεικνύεται. Όλα τα σχετικά με την ασφάλεια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί είναι απλό. Άλλο η ασφάλεια και άλλο η ρήτρα εμπιστευτικότητας. Και είπαμε ότι όλοι οι ετούμενοι θα περνάνε από αυτή τη διαδικασία για την εμπιστευτικότητα, κάτι το οποίο αυτομάτως θα προβλέπεται και υπάρχει ένα δεύτερο μέρος και αυτό θα είναι εμπιστευτικό το οποίο θα αξιολογείται μέσα σε 10 εβδομάδες από την ΕΦΣΑ. το οποίο λέγεται θετικός κατάλογος κριτηρίων και αυτό θα καλυφθεί από την νομοθεσία. Τι θα πει πώς ορίζεται εμπιστευτικό. Εδώ Οπότε η ΕΦΣΑ τώρα θα έχει ξεκάθαρους κανόνες που θα καλύπτουν την πρότασή μας, θα καλύπτονται νομικά Άρα θετική λίστα και το άλλο τμήμα. Και σε 10 εβδομάδες θα υπάρχει ευκαιρία να συλλεγούν πληροφορίες, να γίνει δημοσία διαβούλευση, να αξιολογείται η κατάσταση. Οπότε η ΕΦΣΑ αξιολογεί και αποφασίζει. Αν κάτι δεν είναι εμπιστευτικό μπορεί να το δημοσιοποιήσει η ΕΦΣΑ άμεσα δηλαδή μετά από την περίοδο των 10 εβδομάδων. Επίσης, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η εμπιστευτικότητα κατοχυρώνεται και από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και από το δίκαιο της ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι κάποιοι ειδικοί νόμοι με ειδικέ προϋποθέσεις. Άρα δεν είναι μόνο το γενικό δίκαιο ειδών διατροφής. Άρα θα υπάρχει τώρα ομοιογενής ερμηνεία των κριτηρίων εμπιστευτικότητας. Άρα τώρα θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και θα παράσχουμε εγγύησει για την εποπτεία που πρέπει να υπάρχει από πλευρά κρατική. Και αυτά όλα κατοχυρώνονται από κοινοτική νομοθεσία. Υπολογίζουμε στην βοήθειά σας. Για άλλη μια φορά μπορούσαμε να καταφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα, γιατί θεωρώ ότι η πρότασή μας είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Ούτω ώστε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη εμπιστευτικότητα. Και η κυρία Ρίση μίλησε για τους, αυτούς τους υποκατάστατους συγγραφείς, τους ghostwriters. Ε, το πιο αποτελεσματικό είναι να δίνεται δημοσιότητα και κάποιες εξαιρετικού χαρακτήρα μελέτες της ΕΦΣΑ να μην ε, αποτελούν παρέκκληση και εξαίρεση. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει από την ΕΦΣΑ να αναθέσει μια επιπλέον μελέτη. Και σας ενημερώνω ότι η ΕΦΣΑ αναθέτει, συντάσει πάνω από 400 εκθέσεις το χρόνο. Και βέβαια για τη διφενόλη, για τους διαταράκτες, ε, ε, διάφορα από αυτά που κάνει όπως η Γλυφωσάτη και είναι τον κόσμο οπότε για αυτά ζητούμε εμείς να κάνουν παραπάνω μελέτες να προσλάβουν ειδικού. οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχουν και παραπάνω χρήματα 62,5 εκατομμύρια ετησίες ούτως ώστε να πρικοδοτήσουμε την ΕΦΣΑ και να προσλάβουν παραπάνω κόσμο. 106 παραπάνω είναι αυτοί οι οποίοι προσελήφθησαν λόγω της κοινωνικής χρηματοδότησης. Να μεγάλο βήμα πρόοδο. Έτσι αναβαθμίζουμε την ΕΦΣΑ που μπορούν τώρα να έχουν παραπάνω εμπειρογνώμονες και ειδικού. Κυρία Χάζεκαμπ. Ρωτήσατε για την εμπιστευτικότητα, κυρία Χάζεκαμπ. Τα θέματα αυτά τα έφυξα. Αλλά μιας και μιλάμε για μελέτες, να σας πω ότι τώρα η πρότασή μας επιτρέπει στην ΕΦΣΑ να χρησιμοποιήσει όλα τα επιστημονικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από διαφορετικές πηγές και μελέτες και στη φάση των δημόσιων διαβουλεύσεων υπάρχουν τώρα αρκετές πιθανότητες να λάβει κανείς όλες τις μελέτες που μπορεί να υπάρχουν παγκοσμίω και να τις χρησιμοποιήσει. για την προπαρασκευαστική δουλειά και την ε, προετοιμασία των ε, συζητήσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους. Είναι σημαντική η διαφορά. Έχουμε πολλές συναντήσεις και με μη κυβερνητικές οργανώσεις και αυτές στηρίζουν την ιδέα μας. Θέσατε ένα θέμα για τα εμβόλια και τις διασυνοριακές ζωονόσους. Όταν μιλάμε για διασυνοριακά ζητήματα, δεν είναι το θέμα μόνο μεταφορά των ζώων. Να σας δώσω ένα ε, σημαντικό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ασθένεια η ζωονόσος που ξεκίνησε από την Τουρκία και πέρασε στην Ελλάδα και μετά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πέρασε από κάποιο ζώο αλλά από κάποιο φορέα. Δεν είναι λοιπόν μόνο η μεταφορά των ζώων που είναι υπεύθυνη για την διάδοση ασθενειών. Μερικές τις μεταφέρουν απλώς φορείς. Και δεν αρκεί εμβολιασμό των ζώων. Ε, η πρόβλεψη κάποιων μέτρων. ούτε κάνει μεταφορά των ζώων. Δεν θα μειωθεί επιδημιολογικά η συχνότητα των κρουσμάτων με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το εμπόριο σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών στην ε, Γεωργία. αλλά ε, εμπιστεύομαι και εσά για το πώς μπορεί να ε, βοηθήσετε να βελτιώσουμε τον νόμο. Να ρυθμίσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών καλύτερα με την νομοθεσία και να προβλέψουμε τον εμβολιασμό και για ζωονόσους. Κύριε Χόσλινγκ, θέσατε ερωτήσεις για το πώς εάν δούμε το νομοθετικό πλαίσιο του οργανισμού φαρμάκων ε, και μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτό με ε, την τροφική ασφάλεια. Τα έχουμε συζητήσει αυτά κατά λεπτός, αλλά τα φάρμακα είναι συγκεκριμένα προϊόντα και αγαθό με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε Ε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τόσο διαφορετικά προϊόντα όπως τα φάρμακα με τα τρόφιμα και να προβλέψουμε ανάλογους κανόνες. Έχουμε αξιολογήσει την κατάσταση για τον οργανισμό φαρμάκων, έχουμε συζητήσει για την ΕΚΧΑ. Όλους τους οργανισμούς τον ACDC μαζί και τα βλέπουμε όλα παράλληλα όμως. Η πρότασή μας θεωρούμε ότι είναι και καλά εξισορροπημένη και φιλοδοξή και βοηθά να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, να ανακτήσουμε εμπιστοσύνη και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για την ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης, μιλήσατε για την Επιτροπή των ε, Φυτοφαρμάκων, των Ζανιοκτώνων. Ε, σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για την προστασία των φυτών. Τα θέματα αυτά τα έχω συζητήσει και με τον κύριο Αντριέ και είμαι βεβαίως ότι θα τα καταφέρουμε να τα βελτιώσουμε αυτά προ όφελο των πολιτών μας και να δούμε πως μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά σίγουρα αυτό έχει να κάνει με την προστασία των φυτών και την Περιμένουμε ε, μια αναδιατύπωση που θα ολοκληρωθεί ως το τέλος της χρονιάς. Ε, μια αναδιατύπωση τύπου Refit. Εκεί ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Ε, φυτοφάρμακα ή γλυφοσάτη δεν έχει σημασία. Όλα μαζί θα τα δούμε. Η κυρία Μελάρη ρώτησε για το σύστημα προστασίας των τροφίμων και το πόσο συνεννόμαστε με χώρες που είναι εμπορικοί μας εταίροι, Τρίτε χώρες. Εάν με επιτρέπετε να σας πω ότι τα εμπορικά τα συζητούμε, καθώς και τα φυτο μέτρα, γιατί είναι ε, σημαντικό να ακολουθούνται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν έχουν όλες οι χώρες τα ίδια. Αλλά ένα ευρωπαϊκό προστοποιητικό το παίρνει κάποιο μόνο μετά από εντελεχή έλεγχο και εφόσον έχει προηγηθεί και εκπαίδευση για ασφαλή παραγωγή τροφίμων και χρειάζεται τα συστήματα παραγωγή τροφίμων των χωρών αυτών να ακολουθούν το πρότυπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή δυνατόν να το αντιγράφουν. και να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο ε, ασφάλειας των τροφίμων που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω δεν έχω κάτι να προσθέσω. Απάντησα όλες τις ερωτήσεις. Ναι, Επίτροπε, και πρέπει να περάσουμε και στον δεύτερο γύρο. Ε, ήδη ο πρώτος ήταν πολύ, είπε ο Επίτροπος. Ναι. Τώρα στο δεύτερο γύρο να σας ζητήσω να παραμείνετε στο ένα λεπτό. Η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα επικεντρωθώ στη Γενική Νομοθεσία Περιτροφίμων. Η διαφάνεια, είπατε δύο λόγια και γι' αυτό, αλλά η υποχρέωση δημοσίευσης μελετών. Έχει επιδράσει φυσικά στην γεντομία και στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, αν κάποιος υποχρεωθεί να κοινοποιήσει πιο πολλά δεδομένα από ότι ο ανταγωνιστή του εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Δεν έχει κάνει όμω πανεκτικ τύπου εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και αυτά είναι υποχρεωμένη. Γιατί? Στο 39D του σχεδίου σας αναφέρεται ότι τα πόρτα στοιχεία θα πρέπει να ευδέχονται μετά από αίτημα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. Ε. Όσο εδώ καλά. Αλλά πώ θέλετε, πώς ε, θα διασφαλίσετε να μην υπάρχει διαρροή των απόρριτων αυτών στοιχείων, γιατί φυσικά αυτό εκ νέου αποτελεί α, ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Και άλλη μια ερώτηση, αν θέλετε, για τη δημοσίευση των μελετών, των ερευνών. Αυτό θα ισχύει και για αναδρομικά και στο παρελθόν ή θα ισχύει από την ημέρα της θέσης ισχύς. Ε? Και τι θα γίνει αν παραγωγοί δεν ε, τηρούν αυτά που προβλέπονται. Δεν προβλέπονται κάποιες κυρώσεις και τι γίνεται αν τα στοιχεία αυτά δεν είναι ελέγξιμα και επαληθεύσιμα. Πώς θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν τέτοια στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Καμπεθόν Λουίς. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Να σας πω κάτι για την ψηφιακή υγεία. Ακόμα δεν μπόρεσα να διαβάσω τη χθεσινή σας δημοσίευση, αλλά όπως είπατε θα είναι ενδιαφέρον, έτσι θα βοηθηθούν καλύτερα οι ασθενείς, καλύτερη και η έρευνα θα γίνει, αλλά προβληματίζεται το εξή. Είναι αλήθεια. Είναι σωστό να είναι ο άνθρωπος το επίκεντρο του συστήματος, αλλά να μην ξεχνούμε και τα συστήματα υγείας, τους πάροχους της υγείας. Οπότε αυτή η πρόταση προϋποθέτει καλύτερη διάδοση των δεδομένων. Αυτό θα ωφελήσει και οικονομικά. Αλλά για αυτά τα δεδομένα να μην ξεχνούμε το ότι το κέρδος για τα νοσοκομεία είναι κάτι σημαντικό. Χρειάζεται όλος ο κόσμος να έχει προσβασιμότητα στην υγεία και γι' αυτό σας λέω ότι όσον αφορά την πρότασή σας για την εξατομικευμένη ιατρική κλπ. θα πρέπει να δούμε καλύτερα τις ε, σχέσεις του δημόσιου και του δυτικού τομέα με την έρευνα να υπάρξει το περιθώριο για να βοηθήσουμε τα συστήματα υγείας από οικονομικές. ε, Πάντως η έρευνα θα δώσει λύσεις για όλους τους περισσότερους τέλο πάντων τους Ευρωπαίους που πρέπει να έχουν πρόσβαση ελεύθερη στην υγεία. Η κυρία Κρούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε, για να επανέλθω στο θέμα του εμβολιασμού. Ως γιατρός ε, το ρωτάω αυτό και ξέρω ότι υπάρχουν καινούργιες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλο σε ό,τι αφορά ε, το φράγμα μεταξύ το, του αίματος και του εγκεφάλου. Πάρα πολλά πράγματα είναι ακόμα άγνωστα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα νεογνά, στην εξέλιξη του εγκεφάλου των νεογνών κτλ. Αυτό που θα είχα υπόψη μου ίσως να έπρεπε να απογραφτούν οι εμβολιασμοί τα νεογνά, να ξεκινάνε πιο αργά οι εμβολιασμοί. Ξέρω ότι σε κάποια κράτη-μέλη η θνησιμότητα των ε, νεογέννητων μωρών μειώθηκε δραστικά μετά την απαγόρευση και την, των ε, εμβολιασμών σε νεαρή ηλικία. Κοίτα, θα ήθελα να το εξή. Ε. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών, γιατί υπάρχουν τόσο διαφορετικέ καταστάσει ε, στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη. Κάποια υποχρεωτικά εμβόλια, για παράδειγμα, στην Πολωνία δεν είναι υποχρεωτικά στη δυτική Ευρώπη. Εγώ, για παράδειγμα, δεν βλέπω να υπάρχει σχέση μεταξύ του εμβολιασμού και αντιμικροβιακή αντοχή. Κάποιοι αναφερθήκατε και στα... στην κτηνοτροφία. Δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια σχέση. Η κυρία Ρίζα. Και εγώ για τον εμβολιασμό θα ήθελα να μιλήσω. σε ό,τι αφορά την ε, ανθεκτικότητα στα εμβολιασμό και είμαστε μια και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τον εμβολιασμό, θα ήθελα να πω το εξή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει ένα κείμενο σήμερα το απόγευμα για να δώσει έτσι μια συνέχεια σε αυτή την εβδομάδα. Για παράδειγμα, η κάτι πρέπει να καλυφθεί κατά 95% μέχρι το 2020. Αυτό έχει τεθεί ως στόχο για το 2015. Είχε εγκριθεί αυτός ο στόχος και από ό,τι ξέρετε τα αστικά στοιχεία έχει προκαλέσει ήδη 57 θανάτους το 2017. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν πιο συγκεκριμένα για τα ποσοστά αυτά, για αυτά που αναφέρονται στο σημείο 18 και 19 του ψηφίσματο τη περασμένη Εβδομάδα για το Στρασβούργο σε ό,τι αφορά το θέμα του εμβολιασμού. Ευχαριστώ κύριε Γκέρλινγκ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ένα εισαγωγικό σχόλιο επιτρέψτε μου να κάνω. Όσο Βρετανοί που θα φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πω σε όλου σα να εκτιμάτε αυτά που έχετε. Γιατί με την τρέχουσα νομοθεσία για το τρόφιμα και οποιαδήποτε βελτίωση που ενδεχομένως θα επιέλθει, ε, πρέπει να σας πω ότι εμείς, ε, παρά όλα το γεγονός ότι γκρινιάζαμε ως τώρα, τώρα ανησυχούμε το τι θα γίνει όταν θα σταματήσει να ισχύει αυτή η νομοθεσία, γιατί έχει αποδείξει την αξία τη. Υπάρχουν φυσικά τομεί όπου μπορεί να ε, υπάρξει βελτίωση, επιδέχεται βελτίωση η κατάσταση, αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξει εκ βάθρων να την διαλύσουμε και να την ξαναστήσουμε στα... την πολιτική αυτή. Γιατί την χρηματοδότηση. Μιλήσατε για την αύξηση της χρηματοδότησης με 62 εκατομμύρια. Πείτε μας όμως, αυτό εξαρτάται από το νέο νόμο για τα τρόφιμα, από την νέα νομοθεσία για τα τρόφιμα, μόνο τότε δηλαδή θα διτεθεί. Και πώς θα εγγυηθούμε ότι θα υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση, μήπως ε, θα υπάρξει ένας καινούργιος τελικά νόμος που θα σημαίνει πάρα πολλέ αλλαγέ και θα επιβαρύνει πάρα πολύ και τελικά δεν θα περάσει η χρηματοδότηση. Γιατί φυσικά η διαδικασία είναι εντελώ διαφορετική για την έγκριση τη χρηματοδότηση. Για πείτε μα, λοιπόν, ε, σε τι φάση βρίσκεται η έγκριση τη νέα αυτή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπορζάν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα στην Επιτροπή μα και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τη Γενική Νομοθεσία για το Τρόφιμα και κυρίως για το fitness check. Το περασμένο, το περασμένο καλοκαίρι είχαμε το σκάνδαλο με το φεμπρονίλ, μετά είχαμε την σαλμονέλα στα παιδικά γάλατα το Δεκέμβριο και από ό,τι μας λέει η ΕΦΣΑ, ε, τα κρούσματα σαλμονέλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολλά πολλά χρόνια είναι σε αυξητική πορεία. Όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Οι πολίτες δικαίως ρωτιούνται το σύστημα ασφάλειας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα σωστό στο ύψος των περιστάσεων. Αυτές οι αυτές κάμερα λοιπόν για τα τρόφιμα έληφθησαν ε, υπόψη ε, στις αναλύσεις που έγιναν και τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον ε, για να αποφευχθούν τέτοιες κρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τρίσατε και τον χρόνο, κυρία Αγιούσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον ε, Επίτροπο που ήρθε να μας εξηγήσει τα, των προτάσεων της Επιτροπής. Διάβασα τα της πρότασης νόμου για τα είδη διατροφής. Το θέμα επιδέχεται πολλές βελτιώσεις. Μία από τι βασικέ αρμοδιότητε τη ΕΦΣΑ είναι η αξιολόγηση κινδύνου. Και ισχύει ότι τα φάρμακα είναι άλλη υπόθεση, αλλά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο είδου ε, ε, πιστοποίηση μεταξύ οργανισμού φαρμάκων και διατροφικής ασφάλειας, γιατί δεν είναι ακριβώς ε, το ίδιο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα πρέπει πάντως αυτά τα δύο να βαδίζουν χέρι-χέρι. Τώρα όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις επιχειρήσεις, συμφωνούμε με αυτά που είπε η οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να θέσουν σε εμπορία ένα, κάποιο είδος διατροφής πρέπει να κάνουν έρευνα, πρέπει να επενδύσουν πολλά και οπότε θα πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα την πρόταση ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία όλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι Επίτροπε, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ο κ. Σποκ να κάνει τέτοιες έρευνε και ανανέωση των διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και εκτιμώ την προσπάθεια να γίνει ένα μητρό τέτοιο γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η κατάχρηση των εξαιρέσεων για να αποφύγει κανείς την νομοθεσία. Για παράδειγμα, η προσωρινή απαγόρευση των νέων νοικοτινοειδών. Σε πολλές χώρες δεν πέρασε ποτέ λόγω των ε, εκ της ανάγκης. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και σε όλη την νομοθεσία αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Το ξέρω ότι η ΕΦΣΑ τα εκτιμά αυτή αυτά τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα νεονικοτινοειδή. Αλλά χρειαζόμαστε και μια συστηματική προσέγγιση. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι ολοκληρώθηκε ο κατάλογο ε, των εμπλουτών από τι πολιτικέ ομάδε. Αλλά αν δεν σα πειράζει, έχουμε τρεις συναδέλφους που ήταν εδώ από την αρχή και θα ήθελα να του ακούσω. Η κυρία Σχάιερ Πίρεκ η κυρία Μέλα και η κυρία Ριβασί μετά. Ευχαριστώ πρόεδρε και χαίρομαι που μου δίνετε το λόγο. Το πρόγραμμα εμβολιασμού για το πρόγραμμα εμβολιασμού εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ένα ψήφισμα. Ήταν πάρα πολύ θετικέ οι στην Ολλανδία. Και σήμερα είναι και υπαριθμόν πρώτη είδηση στι συνδέσει, το πώ αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα των εμβολιασμών. Πάρα πολύ θετικό. Να κάνω μια πρόταση. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει και ενημέρωση, πληροφόρηση. Αυτό το είδα και την προηγούμενη εβδομάδα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, τι γίνεται ακριβώς η αντιμικροβιακή αντόχη, γιατί αν δεν καταπολεμήσουμε τα πράγματα στη ρίζα τους, θα ακολουθήσει το επόμενο πρόβλημα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μελέ. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία μελιό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Επίτροπο. Έχω ένα άλλο θέμα να θίξω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους παραγωγούς αρκολούχων ε, ποτών στα πλαίσια της αυτορυθμίσης να καταθέσουν μια πρόταση για τις ετικέτες και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτές. και τη ε, θρεπτική αξία κτλ. Και να δούμε και κάποιες προτάσεις ε, για την επισήμανση και τις ετικέτες. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς όσοι σοσιαλιστές και δημοκράτες θα θέλαμε να υπάρχει και θερμητική ένδειξη, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική συμβολή για την καταπολέμηση ε, της παχυσαρκίας. Η κυρία Τιβασί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει βελτιώσει στη διαφάνεια των μελετών. Αλλά έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο να σας προτείνω, κύριε Ανδρεουκάκης. Γιατί η γλυφωσάτη... ε, 74 μελέτε θεωρήθηκαν εμπιστευτικέ. Αυτό που είναι το πρόβλημα λοιπόν εδώ το εμπορικό απόρριτο. Ή θα πείτε ότι αυτή τη στιγμή οι μελέτε αυτέ έχουν ε, δοθεί στην ΕΦΣΑ και αφορούν ε, τη γενική δημόσια υγεία και ε, προστασία αυτή θα έπρεπε να έχουν δημοσιοποιηθεί. Διότι όταν μιλάμε για τους ερευνητέ, τις εταιρείε και τη χρήση των μελετών τους και χρειάζονται 10 εβδομάδες στην ΕΦΣΑ για να αποφασίσει αν είναι εμπιστευτικέ ή όχι, εδώ έχουμε ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Δηλαδή τι θα πει ότι είναι εμπιστευτικέ πραγματικές μελέτες για το κατά πόσο είναι ασφαλές ένα προϊόν. Δεύτερο, η χρηματοδότηση. Λέτε θα πάρουμε 62,5 ε, εκατομμύρια για να προσλάβουμε τόσους. Μα γιατί δεν πάνε οι μελέτες αυτές στον ίδιο το μηχανικό κλάδο. Και εδώ για τα εμβόλια. Γιατί δεν υπάρχει μία έρευνα ε, για τα εμβόλια, κύριε Ανδρίου για να δούμε πώς μεταβολίζονται τα εμβόλια στον ανθρώπινο οργανισμό. Ε, όλα τα φάρμακα έχουν ε, τέτοιες μελέτες εκτός από τα φάρμακα. Όχι μόνο για τη φαρμακοπαγαπαγρύπνηση λοιπόν, αλλά και για τη φαρμακοδήλη την, του μεταβολισμού τους από τον οργανισμό. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, αν θέλετε έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ε, να απαντήσω στην κυρία Ζόμερ, διότι αναφέρθηκατε στο άρθρο 69D. 39D, με συγχωρείτε. Οι πληροφορίες που ζητήσατε θα διατεθούν στο Ευρωκοινοβούλιο και στα θεσμικά όργανα. Πρέπει ε, επίσης να σεβαστούμε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία και να είμαστε βέβαιοι ότι οι δημοσιεύσεις όλων των εμπιστευτικών στοιχείων πρέπει να ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες. Ως προς τις μελέτες αντεκτύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τα πρότυπα για του κανόνε πνευματική ιδιοκτησία, όπω ορίζονται σε διεθνέ επίπεδο. Η δεύτερη ερώτησή σα αφορούσε το τι γίνεται με τα εργαστήρια που δεν σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να εντοπίσουμε μια ημερομηνία από την οποία και μετά θα πρέπει οι μελέτες να καταγράφονται στο Μητρό. Οι υποχρεώσεις των ετούντων θα πρέπει να μελετώνται από την... Ε, και οι κοινοποίησεις να γίνονται προς την ΕΦΣΑ. Η έλλειψη κοινοποίησης δεν θα... θα πρέπει να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης των ετούντων. γίνονται έλεγχοι και συνεργαζόμαστε και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τα θέματα αυτά. Στην ερώτηση της κυρίας Καμπεζών για την ηλεκτρονική υγεία. Τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε οικουμενική πρόσβαση στο υγειονομικό σύστημα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Και ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αφορά την πρόσβαση στην ε, υγειονομική περίθαλψη. Δεν έχει σχέση ποιος ε, είναι ο ασθενής, αν είναι Γερμανός, Πορτογάλος ή Λιθουανός. Αυτό προβλέπεται με την πρόσφατη πρόσφαση, πρόσβασή μας, οικουμενική πρόσβαση, πρόσβαση για όλου. Κάποιε χώρε αντιτίθενται, αλλά θα δούμε πώ μπορούμε να λύσουμε τα θέματα. Τώρα, στη θέση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Βεβαίω, οι οικονομικέ και κοινωνικέ πτυχέ πρέπει να ε, είναι κάτι που θα το αποφασίζουν τα κρατη μέλη, συμφωνώ. Όμως και η σχέση δημόσια ιδιωτικού τομέα στους πόρους και την παραγωγή των ιατροτεχνικών και το καταξής είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Συμφωνώ. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Πρέπει να το δούμε με πολύ προσεκτικό τρόπο. Χρειάζεται διαφάνεια και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η διαδικασία γίνεται σωστά, ότι το δημόσιο συμφέρον δεν ε, είναι κάτι που, έχει περισσότερη σημασία από τα ωφέλη. Ε, στην κυρία Κρούπα, ως γιατρός για τα εμβόλια, να σας πω ότι με εκπλήσει η ερώτησή σας. Να σας πω τι γίνεται με τι αναλογίε των παιδιών που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αν δείτε τα ιατρικά βιβλία, τα εγχειρίδια της ιατρική. δείτε τα και σκεφτείτε την αξία των εμβολίων. Να δείτε τη σελίδα του ΠΟΗ και τη σελίδα του και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις Νόσους. Υπάρχουν πολλές διαφορε... πολλές σοβαρές διαφορές. Με συγχωρείτε, Επίτροπε, αλλά δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Είπα για την αναβολή των εμβολιασμών μετά το δεύτερο ή τρίτο μήνα. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Δυνατότητες για τον εμβολιασμό νεογνών υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που το συζητάμε εδώ. Πρέπει να συζητηθεί με τους ε, παιδιάτρους, τους ε, ε, ανοσολόγους. Δεν είναι συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα. Υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα στην κάθε χώρα. Άλλες έχουν υποχρεωτικό εμβολιασμό, άλλες όχι. Σίγουρα ζητάμε από τις χώρες να δούμε Ζητάμε από τι χώρε να δουν αυτά τα προγράμματά του και κάποιες φορέ να το προσαρμόσουν. Όμω 70 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν σε διαφορετικές χώρες και ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους από χώρα σε χώρα βλέπουν προβλήματα. Σε κάποιες χώρες ο ε, εμβολιασμό γίνεται πολύ νωρί, ακόμη και στον νεογνά, και σε κάποιες άλλες πολύ αργά. Υπάρχουν ε, δυσκολίες γιατί υπάρχουν διαφορετικά ημερολόγια. Η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με την 20 ε, αιτία. Τώρα επιτρέπεται η κυκλοφορία των ανθρώπων με τις οικογένειές τους. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ε, συμβαδίσουν, να συγχρονίσουν τα ημερολόγια για τον εμβολιασμό, για να προστατεύσουν την υγεία των παιδιών. Και βεβαίως χρειάζονται Και βεβαίω χρειάζονται και φαρμακοκινητικέ μελέτε. Αλλά αυτές οι φαρμακοκινητικές μελέτες ε, από τις υπηρεσίες μου χρειάζονται για όλα τα φάρμακα. Θα το κοιτάξω με τους συνεργάτες μου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω διεξοδικά. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο, θα μπορούσε να γίνει. διότι τα εμβόλια αξιολογούνται πολύ προσεκτικά από τις κλινικές δοκιμές μέχρι την εξουσιοδότηση. Ο έλεγχος είναι διπλός, γίνεται και από τον ΠΟΗ και από τον Οργανισμό Φαρμακών και οι παρενέργειες, όλα. Είναι θέματα που τα παρακολουθούμε κατά προτεραιότητα. Κοιτάμε πώς καταγράφονται, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Έχουμε πολύ ψηλά πρότυπα ασφαλείας για τα εμβόλια και την παραγωγή εμβολίων. Κυρία Ρίσου. ρωτήσατε τι γίνεται με το, παρά, με το της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Τα κράτη-μέλη καταλαβαίνουν ότι ο έχει πολλούς στόχους. Γιατί θέλουμε να υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαλλαγεί εντελώς από τη λαρά στην ουσία αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη. Ντροπή μας που δεν έχουμε απαλλαγή τελείω από την Ιλαρά. Η Βραζιλία ναι, τα έχει καταφέρει και η Πορτογαλία όχι. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε εθνικό επίπεδο τι γίνεται και να αναζητήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Να είμαστε μια ένωση που μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της του ΠΟΗ. Η κυρία Γκέρλι ρώτησε τι γίνεται με τον προπολογισμό. Ο νέο προπολογισμό βασίζεται σε νέα νομοθεσία. Και το τι θα αποφασιστεί και στο πλαίσιο του ποδοπού. Θα πρέπει όμω πρώτα να συμφωνήσετε κι εσείς. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Η κυρία Μπόρζερ ρώτησε γενικώ για τα σκάνδαλα ε, για τα τρόφιμα. Η Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα ε, διασφαλίζει ότι ο νόμος είναι εμ, κατάλληλος για το σκοπό που επιδιώκει. Αλλά όταν μιλάτε για την απάτη, είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε σχέδια δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η κατάσταση σχέση με την απάτη. Υπάρχει και μια μελέτη δικτύπου και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο για την αντιμετώπιση της ε, απάτης στα τρόφιμα, στην παραγωγή τροφίμων και το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο δράσης. Θα σας παρουσιάσω τα πορίσματα της αξιολόγησής μας στο τέλος του καλοκαιριού. Η κυρία Αγιούζο Ε, δεν θα σας δώσω ειδική απάντηση γιατί το κάλυψα με αυτά που είπα στην κυρία Ζόμερ. Σίγουρα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας ε, με περισσότερη λεπτομέρεια σε κάποιες υποθέσεις, αλλά τώρα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες και πώς θα ενισχύσουμε την πρότασή μας. Είμαστε ανοιχτοί στις συζητήσεις με το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο κύριος Ποκ έθεσε θέματα για τις εξαιρέσεις. Σίγουρα εδώ υπάρχουν προκλήσεις και έχουμε διαφορετικές εικόνες στην κάθε χώρα. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχουν χώρες που κάνουν χρήση των εξαιρέσεων με τρόπο ε, τακτικό, οργανωμένο και είναι περίεργο κάποιες φορές να βλέπουμε να τσακώνονται. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση σε διάφορες, στις διάφορες χώρες για να αξιολογήσουμε, να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Αλλά θα δούμε και τι θα γίνει και με το Refit. Και η Επιτροπή θα ε, δει πάλι ε, αν σωστά υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις για να, για να δούμε αν σωστά δίνονται. But, but, but we can cooperate to see how can we move forward. Uh, uh, Madam Schreier-Pirik, okay. Η κυρία Σχαγιοπέρικα, ναι, οι πληροφορίες αυτές ήταν ε, απαραίτητες και συμφωνώ ότι στη νέα πρόταση και στις συστάσεις του Συμβουλίου θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθούν οι εμβολιασμοί. Αυτό θα αποτελέσει ένα καλό βήμα μπροστά, για την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών. Η απάντησή μου είναι ναι, απλή. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις ε, που προβλέπονται από τον νόμο για την θρεπτική αξία, τα συστατικά, τις θερμίδες. Ε, φυσικά και ο, ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται, αλλά τώρα δεν μπορώ να σας πω τι θα προταθεί, γιατί βρισκόμαστε στην φάση της αξιολόγησης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εκπληρωθούν πραγματικά οι διατάξεις του νόμου. Στο έπακρο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τώρα ότι θα πρέπει να γίνουν. Εγώ είμαι σαφώς υπέρ της πληροφόρησης ε, για τα συστατικά, για τις θερμίδες. Ε, δεν ε, βλέπω κανένα λόγο να μην υπάρχουν τέτοιε πληροφορίε. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα τέτοιο λόγο να μην διατυπώνται οι πληροφορίε αυτέ, ό,τι τύπου πληροφορίε και να είναι. Για την κυρία Ριβαζή. Για το κατά πόσο είναι αξιόπιστε οι ερευνέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει τη δυνατότητα να ζητήσει η ΕΦΣΑ έρευνα για την διαδικασία πιστοποίησης. Αυτή η δυνατότητα δεν θα υπήρχε όμως γιατί είναι πάρα πολύ υψηλός ο αριθμός των ετοιμάτων τα οποία κατατίθενται για ε, έγκριση, 450 στον αριθμό περίπου. Και η μεγάλη πλειονότητά τους δεν είναι κάτι το... δεν παρουσιάζει κάτι το αμφιλεγόμενο. Οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο που θα επιλεγόταν το εργαστήριο για την ημερομηνία, την ανεξαρτησία της ΕΨΑ κατά τη διάρκεια των ε, ερευνών και του καθεξής. Και νομίζω ότι έτσι απάντησα στις ερωτήσεις σας. Αν δεν είναι λάθος, η κυρία Σόμερ, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Ζόμερ, μήπω θέλετε να θέσετε εκ νέου το ερώτημά σα. Uh, ναι, Επίτροπε, δεν απάντησα την ερώτησή μου για την ε, έλλειψη μελέτη αντικτύπου για την πρόταση αναθεώρηση του γενικότερου νόμου για τα τρόφιμα. Είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει τέτοιε μελέτε αντικτύπου και ενδεχομένω να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες αν δουλεύουμε στο κενό χωρίς ε, μελέτη αντικτύπου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε μελέτη αντικτύπου. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Τα θέματα αυτά τα συζητάμε. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μελέτης αντικτύπου, καταρχάς για το απόρριτο και την εμπιστευτικότητα δεν χρειάζεται γι' αυτό για θέματα εμπιστευτικότητας και διαφάνειας. Δεν χρειάζεται εκεί μελέτη αντικτύπου. Δεν αφορά κόστος η πρόταση. Μιλάμε για δυνατότητες να αντιμετωπιστούν με σωστό τρόπο α, θέματα που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και με το ρυθμιστικό πλαίσιο, με την εμπιστευτικότητα που θα εφαρμόζονται με σωστό τρόπο. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κενά στην νομοθετική κατάσταση, ότι υπήρχαν ασαφείς καταστάσεις και αυτό δεν προαπαιτεί απαραίτητα διεξαγωγή μελέτης αντικτύπου. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τις απαντήσεις σας. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η ανταλλαγή απόψεων και ο συνήθως με χαρά θα σας προσκαλέσουμε και σε μελλοντικές ε, συναντήσεις μας. Είπατε στην αρχή ότι θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Ναι. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία σας, γιατί σκοπός μας είναι να ολοκληρώσουμε την πρότασή μας σε ό,τι αφορά την ε, τα τρόφιμα μέχρι το 2019. Okay, well, my friends. Uh, uh, να ξεκινήσουμε με το 22 της μερισίας διατάξης που είναι η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, επιλογές σχετικά με τα θέματα της επαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα και απόβλητα. Και να δώσω το λόγο στην κυρία Σχοιερπίρικ η οποία και αντικαθιστά τον συνεισηγητή Λουκάς από το πνεύματα της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, να ξεκινήσω με τα βασικότερα προβλήματα. Ανεπαρκής πληροφορία για ανησυχητικές ουσίες σε προϊόντα και χημικά και απόβλητα. Παρουσία ανησυχητικών ουσιών σε ανακυκλωμένα υλικά θέματα κριτηρίων σε ό,τι αφορά ε, τα απόβλητα, τα οποία δεν θεωρούνται απόβλητα και τέταρτον προβλήματα στην εφαρμογή των διατάξεων για την ταξινόμηση και την κατηγοροποίηση των αποβλήτων και τη διαδικασία ανακύκλωση σε ό,τι αφορά τα δευτερογενή προϊόντα. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα. Και τώρα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον κύριο Λούκα Μάγκλ, ότι βασικότερο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι να αποφεύγει ε, την εισχώρηση επικίνδυνων χημικών στα προϊόντα και για μια σωστή κυκλική οικονομία θα πρέπει να παράγονται προϊόντα τα οποία θα διαρκούν πιο πολύ, θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωή. Και έτσι λοιπόν Η νομοθεσία για τους παραγωγούς και για τα προϊόντα αποτελεί, εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβλημα και μια πρόκληση για τους παραγωγούς. Ε, οι θεμητοί όροι λοιπόν παραγωγής θα πρέπει να εγγυώνται και θα πρέπει τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι σε αρνητική, μειονεκτική μάλλον ε, ανταγωνιστική θέση σε σχέση με τα άλλα προϊόντα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν πιο πολύ συνεργασία και με τα κράτη-μέλη και με την Επιτροπή για τα κριτήρια για το καθεστώ του, γιατί έτσι θα πρέπει να πετύχουμε καλύτερα προϊόντα, τα οποία θα ανακυκλώνονται και θα χρησιμοποιούνται εκ νέου από τους πολίτες. Αυτό θα είναι ε, σημαντικό για όλους. Να δώσω και τη δική μου άποψη θα ήθελα να σας ε, υποδείξω το θέμα του καθορισμού αγρονομικών και περιβαλλοντικών ε, κριτηρίων για τα λοιπάσματα βάσει ε, ζωικών οργανικών ουσιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει όλα αυτά να λεφτήσουν υπόψη και το έχει θέσει και ο κύριος Όγκαν και ο κύριος Τίμερμανς. Επίσης, η κυκλική οικονομία δεν θα μπορέσει να ανακριθεί όσο στην Ευρώπη έχουμε οργανικά ζωικά λοιπάσματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε ως ε, απόβλητα. Και υπάρξει, υπάρχει διακριτική μεταχείριση εν και χημικών ε, λοιπάσματα. Η κατοσαξονία, για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζει την ε, οδηγία για τη μεταφορά των αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα οργανικά λεπάσματα ως απόβλητα. Θέλουμε λοιπόν πιο πολλές οργανικές ουσίες, ε, πιο σωστή επεξεργασία των ε, αποβλήτων. για τη τελική ανάλυση το θέμα είναι να υπάρξει καλύτερη χρήση ξανά και ξανά των πρωτονηλών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για σοσιαλιστές και σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Κάντεμπαχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και μιλώ εξ ονόματος ε, της κυρίας Κρίστελ Κάντεμόζα, η οποία δεν μπορεί να παραβρεθεί εδώ σήμερα, είναι συνεισηγήτρια, αλλά μου ανέθεσε να μεταφέρω τα λόγια της. Το σχέδιο ψηφίσματος που παρουσιάζεται σήμερα έχει ως σκοπό να ε, θίξει πολύ σημαντικέ, αλλά και περίπλοκες ε, λεπτομέρειες και πληροφορίες. Ε. Πιστεύουμε ότι το ψήφισμα, όπως έχει σήμερα, έχει ήδη υψηλό ποσοστό φιλοδοξίας και πιστεύουμε ότι είναι βασικό να αναφέρουμε το εξή ότι ο πιο απλός τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες δεν εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες και χημικά είναι να μην τα βάλουμε στα υλικά και στον κύκλο παραγωγής εξ αρχής. Αυτό θα προστατεύσει την, ευρω... την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά θα διευκολύνει και την μελλοντική γενιά ανακυκλωμένων υλικών και έτσι θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει την κυκλική οικονομία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το θέσει αυτό στόχο υπαριθμών 1 Επίση, για να υπάρξει πλήρη ε, κυκλική οικονομία, αυτό δεν μπορεί να είναι σε βάρο τη ανθρώπινη υγεία και τη υγεία των ζώων και των περιβαλλοντικών προτύπων. Επίση, θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό σκοπό τα προϊόντα σε μια κυκλική οικονομία να έχουν μια μεγάλη διάρκεια ζωή ε, προκειμένου να ε, επαναχρησιμοποιούνται, κυκλώνονται και να επιτερθώνονται εύκολα. Επίση θα πρέπει να αυξηθεί ο όγκος πληροφοριών προς τον καταναλωτή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, γιατί έτσι δεν θα υπάρξει πρόσβαση σε χημικά που δεν θα συνοδεύονται από τι απαραίτητε πληροφορίες. Γιατί αν δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν θα μπορεί να διτεθεί στην εμπορία ένα τέτοιο προϊόν. Θα πρέπει λοιπόν να το θεωρήσουμε αυτό βασικό παράγοντα για την κυκλική οικονομία. Αυτό θα μειώσει και την επιβάρυνση των οικονομικών παραγόντων σε ό,τι αφορά τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που μας ανησυχούν, οι ουσίες που μας ανησυχούν. Έχουμε να πούμε τα εξή. Καταρχάς, πιστεύουμε ότι τα πρωτογενή και τα δευτερογενή πρώτες θα πρέπει να υπάγονται στην νομοθεσία αυτή και οι εξαιρέξεις θα πρέπει να είναι περιορισμένε. Κατά δεύτερον, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της σχετική νομοθεσία στην ευρωπαϊκή αγορά θα βελτιωθεί. Αυτό όχι μόνο για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ όλων, αλλά πολύ πιο σημαντικό στοιχείο για να υπάρχουν τα πιο υψηλά πρότυπα για τον Ευρωπαίο. τέλο. προσβλέπουμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο στις προτάσεις τις οποίες εγκρινάμε χθε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν από το ECR. Ο κ. Κλάρτς από τους Πράσινους. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές δράσεις που έχουν ληφθεί για να έχουμε κυκλική οικονομία για τους πρασινούς αυτό ήταν προτεραιότητα. Ποτέ δεν κάναμε αρκετά για αυτό το θέμα. Και κάθε φόβος είναι δικαιολογημένος και σας θυμίζω τι έγινε με τους διαταράκτες. Στο Άμψεντα συζητήθηκαν οι προσπάθειες βελτίωσης, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα στήματα με κύκλωση. Υπάρχει απαγόρευση από την Κίνα για κάποια πλαστικά και αυτό είναι ευκαιρία για την ανακύκλωση της Ευρώπης και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το θέμα. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάρουν θέση της Κίνας όπως η Μαλαισία και άλλες χώρες. Έχουμε ευθύνη αντί των συμπολιτών μας αλλά και ευθύνη εναντί όλου του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε κυκλική οικονομία ε, όταν ε, τα, τοξικά μας τα εξάγουμε σε τρίτες χώρες. Άρα θα πρέπει με το ψήφισμα να διευκρινίσουμε το ότι θα πρέπει να υπάρχουν εδώ όλες ε, οι ουσίες και όχι μόνο εκείνες που προβλέπονται σε αυτή τη λίστα τοξικά, καρκινογόνα, βιοτοξικά, ε, ανθεκτικά και όλα τα ισοδύναμα. Θα πρέπει να θεωρούνται προβληματικές ουσίες. Και ότι οι ουσίες έχουν ε, επιπτώσεις χρόνιου χαρακτήρα. Υπάρχει ευρωσμική χρήση των πόρων, συμβατότητα, προστασία της ανθρώπινης ε, υγείας και θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα της ανακύκλωσης πέραν των άλλων. Ευχαριστούμε κύριε Σκρίλετς. Γκουέ τώρα. Μπόιλαν. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω μια θετική ανακοίνωση της Κομισιόν όπως και το έγγραφο Εργασίας για τη σχέση μεταξύ των χημικών και της ε, νομοθεσίας για προϊόντα και απόβλητα. Πρέπει όλα αυτά να τα καλύψει η κυκλική νομοθεσία είναι τώρα οι τελευταίες πινελιές, αλλά θα πρέπει, όπως και οι παλιότερες προτάσεις, να λάβουν δημοσιότητα και να ε, προσπαθήσουμε τον ίδιο ενθουσιασμό, όπως και με τα πρώτερα μέτρα. Οπότε θα πρέπει οι πόλεις οι να εξασφαλίσουν ότι η κυκλική οικονομία είναι βιώσιμη και ότι υπάρχει η απαραίτητη νομοθεσία. Γι' αυτό σας λέω ότι χαίρομαι που στο ψήφισμα επισημαίνονται αυτά τα προβλήματα και λέμε ότι θα πρέπει ταχαίως να ενεργήσει η Κομισιόν και η νομοθεσία για προϊόντα, πόβλητα και χημικά να αντιμετωπιστεί σε μια πρόκληση. Άρα θα πρέπει άμεσα αυτά τα θέματα να καλυφθούν. Και όταν μιλούμε για σχεδιασμό, στα πλαίσια της κυκλικής νομοθεσίας θα πρέπει το design των πρέπει να είναι τέτοιο που αυτά να είναι ανακυκλώσιμα και να χρησιμοποιούνται ουσίες που δεν είναι προβληματικές γιατί οι ουσίες τοξικές δεν έχουν θέση στην κυκλική οικονομία. Δεύτερο υλικά επίσης ε, έχουν τοξικές συστατικά, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να επισημανθούν και άρα θα πρέπει έτσι να δούμε πώς θα έχουμε μη τοξικά ε, υλικά όσον αφορά τον κύκλο ζωής τους, να μην έχουμε επικίνδυνα χημικά και κατά δεύτερο λόγο όλες οι προβληματικές ουσίες θα πρέπει να ανοιχνεύονται και θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενημέρωση προς ανακυκλωτές και προς το κοινό. Τα απόβλητα θα γίνονται πρωτήλοι και οπότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν, όλα αυτά αποτελούν προβλήματα για το μέλλον. Τέτοια στρατηγική θα πρέπει να συνεχίσουμε να την προσέχουμε όσον αφορά την χρήση εκμετωσή προϊόντων όσο λιγότερο πλαστικό χρησιμοποιούμε, τόσο πιο εύκολο θα λύσουμε το πρόβλημα για αυτή τη σχέση της νομοθεσίας με τα τοξικά και με ε, τα πλαστικά το οποία προβλήματα για το απότερο μέλλον. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε τους συνεισηγητές. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. κυρία ε, και πρόεδρε, ένα σημείο που ξέχασα Πρωτού πάρω το λόγο οι συνάδελφοι για τη συζήτηση στο Άμστερνταμ. Θα θέλαμε να πούμε το εξή, ότι λάβαμε παραπληκτικέ προτάσει από εταιρείε και ανθρώπου που προσπαθούν να παράγουν δίζελ από πλαστικό και σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν λαμβάνουμε τόσες πολλές προτάσεις που είναι εντυπωσιακό. Θα πρέπει κάτι να τις αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν βλέπω και κανέναν άλλο να παίρνει το λόγο. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που βάλετε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Όπως είπε και η εκπρόσωπο τη ΕΕ, αυτή η πρόταση μπορεί να μην έχει λάβει την ε, προσοχή που έλαβε η πρόταση των πλαστικών τότε, αλλά να σας πω ότι είναι εξίσου σημαντική. Γιατί αν δεν το πετύχουμε αυτό, δεν θα υπάρχει κυκλική οικονομία. Ας δούμε λοιπόν το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που προτάθηκε το 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι οι στόχοι που είχαν προταθεί τότε εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ επίκαιροι εδώ. Για παράδειγμα, η κυκλική οικονομία, ένα μοντέλο όπου διατηρείται η αξία ενός προϊόντος μιας ουσίας όσο πιο πολύ γίνεται, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την άσκηση αυτή διαπαθής. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να διτηρηθεί η αξία, σε περίπτωση που ε, ένα προϊόν ε, είναι ανεπιθύμητο λόγω παρουσίας α, επικίνδυνων ουσιών που αποκαλύπτεται όταν το προϊόν είναι ακόμα στην αγορά ή, για παράδειγμα, μπορεί να περιοριστεί η ανακυκλισμότητα αν μιλάμε για επικίνδυνες ουσίες ε, στο προϊόν ακόμα χειρότερο, άμα δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτή η ουσία, δεν είναι γνωστή η σύνθεση του προϊόντος και γίνεται ανακύκλωση του προϊόντος σε κάποιες περιπτώσεις και αυτό το αναφέρουμε και στο σχέδιο δράσης δεν είναι τα συμφέροντα των ε, παραγωγών στην αλυσίδα παραγωγή. Ε, σε κάποιε περιπτώσει ε, συνάδουν βέβαια. Θα πρέπει να βρούμε εδώ λοιπόν μια ισορροπία. Και ακριβώ αυτή την ισορροπία επιδιώκουμε να πετύχουμε. Στην ανακοίνωση και στο έγγραφό μα έχουμε δώσει πολλά παραδείγματα για το πού ενδεχόμενες τέτοιες ε, διαφορετικές ε, συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να εντοπιστούν και πού θα πρέπει να λεφθούν αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις και ε, μπορεί να είναι παραδόξως το να επιτρέψουμε σε κάποια προϊόντα και κάποιες ουσίες να χρησιμοποιούνται ακόμα για να διατηρηθούν κάποια προϊόντα. Και νομίζω ότι στην Επιτροπή μας είχαμε συζητήσει την ε, ε, οδηγία ΡΟΖ για τα ηλεκτρονικά και τα επικίνδυνες ουσίες ηλεκτρονικά. Εκεί λοιπόν απο... επιτρέψαμε κάποιε ουσίε να περιλαμβάνονται σε κάποια εξαρτήματα προκειμένου κάποια προϊόντα όπως για παράδειγμα ηλεκτρικά ποδήλατα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, και στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να κυκλοθούν. Δεν το επιθυμούμε αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε και να ερευνήσουμε με ευρύτερο τρόπο όλες αυτές τι αποφάσει που θα πρέπει να λεφθούν. Κάποια από τα στοιχεία έχουν ήδη ε, εκτελεστεί για τη Γερός, για παράδειγμα. Επίσης, η Επιτροπή σας δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την, τα απόβλητα. Πολύ καλέ διατάξει περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι διατάξει ε, για την απολύμανση. για παράδειγμα, οι διατάξει για την ειχνηλάτηση των ουσιών. Σε ό,τι αφορά ουσίε ε, που μα ανησυχούν ιδιαίτερα, οι οποίε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΡΙΤΣ, αλλά και με συγκεκριμένο, δομημένο τρόπο, προκειμένου να δίνονται αυτές οι πληροφορίε τελικά στους ε, αρμόδιους Ύστερα, σε ό,τι αφορά την ε, ταξινόμηση των αποβλήτων, τέταρτο στόχο, πριν από κάποιε εβδομάδε δημοσίευσαμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ λεπτομερεί κατευθυντήριε γραμμέ για την ε, ταξινόμηση των ε, αποβλήτων. Γιατί και εδώ υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει μεταξύ κρατών μελών. Κάποιοι τα θεωρούν επικίνδυνα, κάποια απόβλητα, κάποια άλλοι όχι. Πώ τελικά οι υπεύθυνοι θα τα κατατάξουν, θα τα στείλουν, θα τα μεταχειριστούν τα απόβλητα αυτά. Είναι πολύ ε, σαφείς και απτές προκλήσεις και δυσκολίες, ε, τις οποίες ε, μας, τις μας την επεσήμαναν στις διαβουλεύσεις ε, η κοινωνία των πολιτών, οι εμπλεκόμενοι φορείς, μας είπαν, κοιτάξτε, αυτά μας απασχολούν, αυτά είναι τα πραγματικά θέματα που θα πρέπει να επιλύσουμε. Γι' αυτό και σε αυτά επικρινόμαστε. Θα πάρει κάποιο χρόνο, δεν μπορεί. Και είναι και μια διαδικασία εξισορρόπησης, μην αμφιβάλλετε αλλά φυσικά και προσβλέπουμε στις εργασίες αυτές τους επόμενους 24 μήνες, λίγο πολύ, γιατί είχαμε πει ότι θα βρούμε λύσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα αναζητήσουμε λύσεις μέχρι το τέλος του 2019. Θα χρειαστούμε καθοδήγηση και από δική σα πλευρά. Και γι' αυτό λοιπόν το ψήφισμα είναι πολύ επικοδομητικό. Το καλωσορίζω το ψήφισμα αυτό θα το δούμε και τον θα έχει ε, εγκριθεί, μία μικρή πρόταση, αν τρέπετε. Όταν ε, απαριθμείτε διεθνείς ε, συμβάσεις όπως το για παράδειγμα, ή της Βασιλείας, να αναφέρετε και την σύμβαση του Σόγκολ για την παρουσία ρηπαντών. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και φυσικά θα χαρώ να συνεργαστούμε για το θέμα αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Δίκη Πρόεδρο. Για το χρονοδιάγραμμα 2 Μαΐου η υποβολή τροπολογιών στις 11 το πρωί θα ψηφιστεί στην Επιτροπή ΕΜΒ 21 Ιουνίου και στην Ολομέλεια κατά πέσα πιθανότητα τον Ιούλιο φέτος. Ξεκινάμε τώρα με το σημείο 23 στην ημερήσια διάταξη. Προστασία της εσωτερικής αγοράς και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου, της παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς. Υπάρχει κάποιος από το έλεγχο που να αντικαθιστά την κυρία Ζόμερ. Όχι από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες εγώ, οπότε θα περάσω στα τσεχικά. Το παράνομο εμπόριο των ζώων συντροφιά είναι ένα ε, φαινόμενο που δεν αντιμετωπίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές καταχρήσεις σε πολλά κατημέλη, όπως στην ε, Δημοκρατία της Τσεχίας, όπου για την εμπορία γατιών, σκυλιών είναι πολύ χαμηλά τα πρότυπα. Πολλές ε, φορές παρακάμπτεται η οδηγία 92 και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα εμβόλια. Απειλή για την δημόσια υγεία και παραπλάνηση των καταναλωτών είναι τα αποτελέσματα. Επίσης υπάρχουν ε, ε, κέντρα αναπαραγωγής τα οποία είναι παράνομα και ε, παράνομο εμπόριο στο διαδίκτυο. Δηλαδή μπορεί να κερδίσουν εκατομμύρια τσεχικές κορώνες οι παράνομοι έμποροι. Παραποιούν τα έγγραφα των ζώων και τα ζώα, τα νερά ζώα, μεταφέρονται σε πολύ αρνητικές συνθήκες. Συνθήκες που υποβαθμίζουν την υγεία τους. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κατημέλη να κάνουν τα εξή. Πρώτα απ' όλα, να εντοπίσουν και να καταγράφουν σωστά τους σκύλους και τις γάτες που θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα στην καταπολέμηση με το παράνομο εμπορίου. Δεύτερον, να δημιουργήσουν μια διεπιστημονική γραμμή δράση για να αναλάβουν την ευθύνη όλοι οι αρμόδιοι ε, φορεί και μετά να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ 100 μελών για να επιληθεί εν τέλει αυτό το πρόβλημα. Να ευχαριστήσω τι τσεχικέ με κυβερνητικέ οργανώσει για τη συνεργασία του τη Λίγκα για την προστασία των ζώων, το Animal Eye και, άλλα, ε, ε, και άλλες ενώσεις όπως την Dog Trust. Τώρα, ο κύριος Εκ από την Γκουε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, και για τη δική σας εισήγηση. Δυστυχώς η πώληση γνώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστιο ε, ένα τομέα που δίνει τεράστια κέρδη με πολλού ε, παρανομούντε να εμπλέκονται εδώ. Τα ζώα αναπαράγονται εκτός ε, νομίμων συνθήκων. και μεγαλώνουν σε συνθήκες ε, ανθυγιεινές. Δεν εμβολιάζονται και όπως λέτε και το διαδίκτυο συμβάλλει στη διόγκωση αυτού του εμπορίου. Είναι τέλεια πλατφόρμα για να κάνει κανείς ε, να αποκομίσει κέρδη εκατομμυρίων χωρίς να πληρώνει φόρους. Η λοιπόν προβλέπει να ε, υπάρχει καταχώρηση όλων αυτών των ε, παραγόντων, αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλά κενά και γι' αυτό πολλά παραθυράκια χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ε, μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια σε ό,τι αφορά του εμπόρου ζώων. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των εγκληματιών αυτών, σε ό,τι αφορά την εμπορία τέτοιων των, των ζώων. Θα πρέπει λοιπόν ε, τέτοια συστήματα και μητρώα προκειμένου να ελέγχεται η ταυτότητα των ατόμων αυτών και των εκτροφέων ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ρυθμιστούν όλα αυτά σε ό,τι αφορά την εκτροφή. Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, αθέμητες πρακτικές εμπορίου και τα τα ουσιαστικά των ζώων. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να πάρουμε αυτά ένα τέρμα. Σας ευχαριστώ. Από το Διευθυντή, η κυρία Ρίτ. Pleasures. Uh, Προφανώς είναι πρόβλημα αυτό. και, το, και η ομάδα μου δεν θα ήθελε να φτάσει στην έσχατη λύση των διαπιτηρητήριων για ζώα των διαβατηρίων για ζώα. Αλλά πρέπει κυρίως να δούμε για τους εμπόρους αυτών των ζώων συντροφιάς ε, τι νομιμοποίηση θα λαμβάνουν, πώς θα ελέγχονται και πώς θα καταγράφονται σε κάποιο μητρό. Έχουν την σωστή άδεια. Υπάρχει τρόπος ε, το κάτω να ξέρει ότι μπορούν να ε, οργανώνουν την αναπαραγωγή των ζώων. Γιατί και τα ζώα έχουν δικαίωμα να είναι υγιή. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν να προβλέψουν αυτές τις ε, εγγύησει. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς όχι. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Φίσιλ από την DG Σάνκο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αυτή τη στιγμή ασχολόμαστε με την υλοποίηση της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς που εγκρίνατε εσείς και το Συμβούλιο στις 9 Μαρτίου 2016. Τελική ημερομηνία ήταν ο Απρίλιος 2021 όπου όλες οι νέες διατάξεις θα έπρεπε να ισχύουν. Βεβαίως, η νομοθεσία για την υγεία των ζώων προβλέπει περισσότερες δυνατότητες από την τωρινή νομοθεσία, η οποία βασίζεται σε οδηγίες και πιο πρόσφατα κανονισμό. Αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερο το Κοινοβούλιο, εισήγαγε συγκεκριμένες γραμμές για τα ζώα συντροφιάς, γιατί το άρθρο 277 της ε, νομοθεσίας για τα ζώα και την υγεία των ζώων λέει ότι οι τωρινοί κανόνες για τη μη εμπορική μεταφορά των ζώων συντροφιάς πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το 2026. Προς στιγμή, λοιπόν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο προτεραιοτήτων μας. Το 2019 είναι οι πρώτες προθεσμίες μας γι' αυτό και όχι το 2026. Και σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγή και την καταγραφή των ζώων, βεβαίως η νομοθεσία για την υγεία των ζώων ανοίγει νέες δυνατότητες και επιτρέπει να διευρυνθεί η υποχρέωση καταγραφής των κέντρων αυτών που ασχολούνται ε, με την αναπαραγωγή ενδοευρωπαϊκά για εμπορικού σκοπούς. Παραμένει όμως το πρόβλημα της δυσκολίας να ανοιχνεύσουμε όλα τα νοικοκυριά, τα ιδιωτικά νοικοκυριά που αποκλείονται ε, συγκεκριμένα από αυτές τις υποχρεώσεις ε, καταγραφής από την νομοθεσία. Είναι ένας χώρος αχαρτογράφητος. Είναι δύσκολο το εντάξουμε στην υγεία των ζώων τώρα τις ε, επιγραμμικές πωλήσει και τους σχετικούς κανόνες, αυτό είναι διαφορετικό. Να σας θυμίσω ότι επίσης έχουμε το νέο κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους που εξετάζει το θέμα της υλοποίησης και βάσει αυτού Ζητούμε τις καθεξουσιοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να διεξαγάγουν τους ε, απαραίτητους ε, ελέγχους για, την, ε, για τις επιγραμμικές πωλήσει και τη συμμόρφωσή τους με τους νόμους. Δεν μπορώ να είμαι πιο λεπτομερής από τευτό. Δεν μπορούμε να, επανα, να επανεφεύρουμε υπάρχοντε κανονισμού. Βεβαίω τα κάτι μέλη έχουν υποχρεώσει που απορρέουν από όσα ισχύουν για το εμπόριο. Αλλά ζήτησα από του συναδέλφου στην DigiTrade να μου δώσουν μια σύντομη συνοπτική εικόνα για το θέμα αυτό. Και σίγουρα υπάρχει σήμερα παράνομο εμπόριο, αλλά Υπάρχουν και ένα εκατομμύριο ζώα που είναι αντικείμενο εμπορία τα τελευταία πενταετία. Πλήρω συμμορφούμενα με την πιστοποίηση και όσο απαιτείται για το αρχείο, το μητρό, την καταγραφή των κινήσεών τους αλλά υπάρχει και ένας τομέας χώρος όπου δεν έχουμε γνώση για την πρωτογενή κυκλοφορία των ζώων. Ε, είναι λίγο δύσκολο να πιάσουμε τα νοικοκυριά που κάνουν και εμπόριο. Χρειάζεται πολλή εκπαίδευση των πολιτών για να καταλάβουν τι ευθύνη να αναλαμβάνουν όταν ε, παίρνουν ένα ζώο, το ζώο δεν είναι κάτι που το πετάς μόλις βαρεθείς. Αν δεν είναι πολύ και όσο ενθουσιασμός που το πήρες. Νομίζω ότι την πλευρά μας όμως είμαστε όσο πιο δραστήριοι γίνεται και έχουμε την κατάλληλη νομική βάση για να ε, υλοποιήσουμε και να ελέγξουμε αυτό το είδο το εμπόριο. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Α, ήρθε η κυρία Ζόμερ. Φαντάζομαι ότι θέλει να λάβει το λόγο. Και τη τον δίνω. Ευχαριστώ πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσα. Σήμερα το πρωί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη γιατί έχουμε και την αντιπροσωπεία με την Τουρκία και έχουμε και Τούρκου ομολόγου μα μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ήρθα επιτέλου. Και διάβασα και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σα επενθυμίσω ότι είχαμε ήδη ένα ψήφισμα τον Φεβρουάριο του 2016 για το θέμα αυτό. Δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε θέματα υγείας των ζώων. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της υγείας των ζώων για την, ευρωπαϊκό, για ευρωπαϊκή διάσταση σε ό,τι αφορά και τα κρατημέλη τα οποία μπλοκάρουν, για παράδειγμα, πολλή νομοθεσία. Αυτό που προγραμμίσαμε όμως ήταν το εξή ότι δεν αποτελεί αυτό μόνο πρόβλημα της υγείας των ζώων και της ευημερίας των ζώων. Τίθεται και θέμα μαζικά για τη δημόσια υγεία την ανθρώπινη υγεία, γιατί αυτό το παράνομο εμπόριο οικιακών ζώων θετει και θέματα διεθνή εγκληματικότητα, εγκληματικότητας και Δημόσια υγείας. Μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη πηγή προσόδων μετά το παράνομο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Πώ μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό και τίθεται και θέμα ιστορική αγορά. γιατί φυσικά μαζικά υπάρχει και φόρο διαφυγή. Μετά στο ψήφισμά μα λοιπόν πριν από δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δραστηριοποιήθηκε την για θέμα αυτό και το βέτο λοιπόν εκ νέου. Είναι επικίνδυνο για τον κόσμο να έχει ζώα, για παράδειγμα, τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί, χωρίς να το ξέρει, ε, που είναι νοσούν χωρίς να το ξέρει ο διευθυντής της. Ή να χάνεται το, η ζωή του ζώου, να χάνεται το ίδιο το ζώο και να έχει πληρώσει και ένα σκασμό λεφτά για ράτες οι οποίες δεν χρειάζεται να πληρώσουν. Πάρα πολλά λοιπόν μπορούν να μεταφερθούν και προς τον άνθρωπο. Πολλές είναι οι που επηρεάζουν και την ανθρώπινη υγεία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και όλα αυτά που έχουν γίνει ως τώρα και η αναθεώρηση του διαβατηρίου των ζώων. Ούτε αυτό βοήθησε. Θα πρέπει επιτελούς να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό προφανώς είναι στα χέρια της Γενικής Διεύθυνσης ε, Υγείας ε, DG Santa. Μιλάμε για θέματα δημόσιας υγείας. Και να επιθυμήσω στους αδέλφους το εξή. Στο σχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας, και για το οποίο θα καταθέσουμε ε, τροπολογίες μέχρι την άλλη εβδομάδα από την Νομίζω ότι πολλά συγχαίουμε. Καταρχάς όταν μιλάμε για τα ζώα συντροφιά. Μιλάμε για σκύλες, και γάτες. Δεν είναι χελώνες και φίδια. Μην ε, προκαλείται λοιπόν σύγχυση μεταξύ των κατοικιδίων και των ζώων συντροφιά. Είναι κάτι διαφορετικό. Και ανησυχώ, ανησυχώ λίγο σε ό,τι αφορά το νέο αυτό ψήφισμα. Να προσέξουμε, να μην αποδυναμώσουμε το προηγούμενο ψήφισμα. Θα πρέπει να κάτσουμε σε να συζητήσουμε. Θέλω να βελτιάσω την κατάσταση. Προφανώς και εγώ θέλω και τα άλλα ζώα. Τα οποία βρίσκονται στα νοικοκυριά χωρίς λόγο σε διάφορες περιπτώσεις όταν πρόκειται για ρηπετά και άλλα είδη. Και για αυτά λοιπόν τα ζώα θέλω να κάνω κάτι, γιατί πραγματικά ε, είναι βασανιστήρια για τα ζώα αυτά. Χωρίς να το ξέρει και το καταναλωτή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδυναμώσουμε την ε, νομοθεσία για τα ζώα στροφιάς. Να επισημάνουμε εκ νέων αυτά που είχαμε αποφασίσει πριν από δύο χρόνια και όχι να μειώσουμε την ισχύ αυτών των διδάξεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. Για τις ε, τροπολογίες είναι Δευτέρα Μαΐου, καταληκτική ημερομηνία. Και 21η Ιουνίου θα ψηφίσουμε και θα πάει μάλλον στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Δεν έχουμε κάτι τίποτα διάφορα. Απλώς σας ενημερώνω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει 16 και 17 Μαΐου. Καλό απόγευμα. Γεια σας.